Okay, colleagues. Καλώς ήλθατε αγαπητές και αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Είναι βέβαια απόγευμα, αρχίζουμε με κάποια καθυστέρηση. Αλλά έχουμε φτάσει 3 και 10. Έχουμε και συναδέλφους από πολλές πολιτικές ομάδες. Έχουμε ήδη ένα αριθμό συναδέλφων παρούσες και παρόντες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη συνεδρίαση του 2016. Έχω ήδη συναντήσει κάποιους από εσάς στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και πάντως εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά. Θα έχουμε και τον Επίτροπο με μέλη του γραφείου του και ελπίζω να είναι επιτυχημένη αυτή η αρχή του 2016, η πρώτη αυτή συνεδρίαση. Θα δεχτούμε επίσκεψη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής ε, των Κοινοτήτων για τη διεθνή ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας για να κάνει τις συστάσεις. Μετά θα πάνε στα ξενοδοχεία τους και θα επανέλθουν στη διάρκεια της συνεδριάσεως. Πρώτα λοιπόν για το υπαριθμόν 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως δεν έχουμε αλλαγές ή μάλλον έχουμε μία αλλαγή, συγγνώμη, ο Brian Hayes που έχει αναλάβει τη γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον έχει άλλη υποχρέωση σε άλλη ε, κοινοβουλευτική επιτροπή και γι' αυτό ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε το υπαριθμόν 9 θέμα να το συζητήσουμε πριν από τα 7 και 8. Αυτό είναι το δικό του θέμα δηλαδή. Δέχεστε να εγκρίνουμε την μεσία διάταξη με αυτή τη μικρή αλλαγή. Σας ευχαριστώ λοιπόν. το υπαριθμόν 2 ανακοινώσει της Προέδρου. Ήδη έκανα μία από τις ανακοινώσει αυτές, ενώ την επίσκεψη της Επιτροπής τη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεύτερη, μετά από απόφαση των συντονιστών, το Policy Department έχει οργανώσει ένα εργαστήριο για την συνοχή της πολιτικής της αναπτύξεως με τίτλο «Ευρωπαϊκή πολιτική μάλλον συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη και η πρόκληση της ε, βιωσιμότητας, στα οποία θα συμμετάσχουν και ομιλητέ από τον ΟΣΑ, UNDP και θα γίνουν στις 16 Φεβρουαρίου, εκτός ορών της ε, εργασίας της Επιτροπής μας. Ξαναλέω, στις 16 Φεβρουαρίου, στις 12.30 στην παρούσα αίθουσα. Ελπίζω να μπορέσετε να είστε παρούσες και παρόντες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πολιτική αυτή. Και αυτή η πολιτική είναι εκείνη που ξεχωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Δηλαδή φροντίζουμε όσα γίνονται, όσα κάνουμε σε ορισμένους τομείς πολιτικής να μην έρχονται σε αντίφαση με άλλα. Ο κ. Πέντερ θα είναι ο εισηγητής, θα αναλάβει την έκθεση. Ελπίζω να έρθετε στο εργαστήρι αυτό. Οι δε συντονιστές των πολιτικών ομάδων να υπενθυμίσουν το ε, εργαστήριο αυτό στα μέλη των ομάδων τους. Ας καθίσουν τα μέλη της ε, Βουλής των Κοινοτήτων και μετά θα σας δώσω το λόγο κύριε Πρόεδρε για να μπορέσετε να ε, κάνετε τις συστάσεις. Αν θέλετε να πάρετε νερό ή βρίσκεται εκεί. Είναι do it yourself εδώ το νερό. Το υπαριθμό 3 είναι έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδριάσεως που ήταν 20 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2015. Τα έχετε στους φακέλους σας. Αν έχετε παρατηρήσει σχετικά με τα πρακτικά να ενημερώσετε τη γραμματεία της Επιτροπής πριν από το τέλος της συνεδριάσεως. Και αν δεν λάβουμε τέτοια σχόλια θα θεωρήσουμε ότι τα εν λόγω πρακτικά εγκρίνονται. Αυτά για το υπαριθμό 3. Υπαριθμό 4. Ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι παρούσα βεβαίω. Δεν ξέρω αν οι υπηρεσίε τη Επιτροπή έχουν κάποιε ανακοινώσει τι οποίε επιθυμούν να προβούν. Όχι. Τίποτε. Πάντω είστε παρούσα. Αλλά δεν πρόκειται να προβείτε σε ανακοίνωση. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Εάν ο Στίβεν Τρίγκ που είναι επικεφαλής της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων για θέματα διεθνούς αναπτύξεως βεβαίω αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνεργαζόμαστε σε πολλά ε, σχετικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι εσείς αναλάβατε πρόεδρο τον Ιούλιο. Η δική μα επιτροπή είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη ειδική από τη δική σα. Στίβαν, θέλετε να κάνετε τι συστάσει ε, τη Επιτροπής. Λίντα, σα ευχαριστώ πολύ. Και καλησπέρα σε όλε και όλου. Με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε εδώ. Λέγομαι Steven Twig Είμαι των εργατικών, μέλος ε, της Βουλής των Κοινοτήτων από το Ενωμένο Βασίλειο. Είμαστε διακομματική επιτροπή από όλα τα κόμματα δηλαδή και αυτό που κάνουμε είναι ασκούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο ε, Υπουργείο Περιφερειακής Αναπτύξεως. Και ε, όπως είπες Λίντα ανέλαβα την Προεδρία των Περασμένου Ιούλη για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των ε, θεμάτων της ανάπτυξη. Ως Επιτροπή λοιπόν μα ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία ε, ημών ω Εθνικής κοινοβουλευτική επιτροπή, με τη δική σας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διήμερης επισκέψεως. Θα συναντήσουμε ορισμένε και ορισμένους εξημών ανεπισήμως αργότερα. Έχουμε πολλές ε, συναντήσεις και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μας ε, ε, δίνετε την ευκαιρία να είμαστε εδώ και αναμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε τις συζητήσεις σας. Dear Νέβα, ίσως αργότερα. Πολύ καλώ. ήλθατε. Είχαμε επίσκεψη την προηγούμενη, μάλλον στις αρχές του χρόνου, από την γερμανική Bundestag συναντηθήκαμε και στο Λουξεμβούργο υπό την διεύθυνση της Λουξεμβουργικής Προεδρίας βουλευτών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, τη διεθνή ανάπτυξη, πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία αυτή. Στο τέλος τη συνεδριάσεω μα, στι 6.30 δηλαδή, γιατί οι συνάδελφοί μα από το Ενωμένο Βασίλειο θα μεταβούν και σε άλλε επιτροπέ, αλλά πάντω στι 6.30 θα επανέλθουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε έναν ανεπίσημο διάλογο με ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες μέλη και διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες. Είστε λοιπόν εγκάρδια προσκεκλημένες και προσκεκλημένοι όλοι εδώ για να συζητήσουμε και μετά θα έχουμε και ένα ποτό. Αν λοιπόν είστε διαθέσιμοι, ελάτε να μπορέσετε να συνομιλήσετε με τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων. Καλώς λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα στην παριθμόν 5 της ημερησίας διατάξεως. Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως και το εργαλείο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Θα προβούμε σε διάλογο με τον ε, Επίτροπο Νέβεν Μίμητσα. Χαίρομαι πολύ κύριε Επίτροπε που είστε παρόν τώρα στην πρώτη μας συνάντηση του 2016. Ε, βεβαίως εδώ λίγη η πρώτη σας χρονιά ως ε, Επιτρόπου αλλά και η δική μας ως Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο περσινός χρόνος ήταν σημαντικός. Ήταν ε, το έτος της αναπτύξεως, ευρωπαϊκό έτος αναπτύξεως, αλλά και σημαντικών συμφωνιών, καθώς και της ατζέντα για τα επόμενα 15 χρόνια. Έχουμε λοιπόν συμφωνία για τις SDG στη Νέα Υόρκη με ε, προσώπους και από εσά ε, για την Βέμπα, για, στην Βέμπα μάλλον για την χρηματοδότηση και στο Παρίσι βεβαίως η Μεγάλη Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που ασφαλώς και αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ατζέντα για την ανάπτυξη. Είναι και ο πρώτος χρόνος για το νέο αυτό εργαλείο της συνεργασίας για την ανάπτυξη που πηγαίνει μέχρι το 2020, 2014-2020 και τα ίδια τα προγράμματα αυτά είχαν ε, συμφωνηθεί και εγκριθεί από το προηγούμενο Ευρωκοινοβούλιο 14-19. Για ορισμένα όμως μέλη μας είναι νέα προγράμματα αυτά. Δεν είχαμε ασχοληθεί με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, καλούμεθα όμως να τα εφαρμόσουμε. Αλλαγέ έγιναν επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή διαθρώνονται οι υπηρεσίε τη. Τώρα έχουμε, είπα το εκπρόσωπο που προεδρεύει όλων των συναρμόδιων επιτρόπων ώστε να υπάρχει συνοχή στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική διεθνού ανάπτυξη. Έχουμε και καλύτερη συνεργασία στον προγραμματισμό μεταξύ χωρών μελών και μεταξύ του αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινούμε λοιπόν μια νέα εξαετή περίοδο της ε, πολιτικής αναπτύξεως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει τον ρόλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ε, πολιτικής αναπτύξεως. Περάσαμε ένα χρόνο για να μάθουμε λίγο πώς λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε πέντε ομάδες εργασίας που ε, ασχολούνται με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και που προβαίνουν σε διάλογο όπως προβλέπει το εργαλείο της συνεργασίας για την ανάπτυξη έχουν πολυενδεικτικά προγράμματα, προγράμματα δράσεων και ειδικά μέτρα. Ασχολούμεθα και με τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και οι συνάδελφοι ενώ και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι έχουμε δύο τρόπους χρηματοδοτήσεως. Έχουμε χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού όπου εκεί εμείς είμαστε αρμόδιοι για την εποπτεία του DCI, του εργαλείου δηλαδή για την ε, συνεργασία στην ανάπτυξη, και για τις χώρες ε, που βρίσκονται στην πορεία της ένταξης και τις γειτονικές τους. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό βέβαια Ταμείο Αναπτύξεως. Διμερές ε, ταμείο στο οποίο καταβάλουν σφορές οι κυβερνήσεις και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τις χώρες Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού στη βάση της Συμφωνίας Κοτονού. Και θα δούμε εάν αυτό θα διατηρηθεί το πλαίσιο αυτό ή αν θα αντικατασταθεί από νέο. Πάντως αυτά είναι τα νέα προγράμματα. Τέλος, την προηγουμένη εβδομάδα συναντήθηκαν οι συντονιστές μας για να συζητήσουν πώς ε, εφαρμόζεται ο κοινοβουλευτικό μα έλεγχο. Έχουμε καταθέσει ορισμένε ιδέε για την βελτίωση του δικού μα ρόλου. Έχουμε ορισμένα πράγματα που θέλουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, κύριε Επίτροπε, θα δώσω πρώτα το λόγο σε εσά και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη μα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Λίντα, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή, για τα καλά σας λόγια και προσβλέπω στην συνεργασία μας κατά τη διάρκεια του 2016 να ξεκινήσουμε ε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τα πιο σημαντικά και πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Σωστά αναφέρατε ότι είχαν τη σημασία των διασκέψεων στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Ναϊρόμπι. Έγιναν όλες αυτές οι εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο. Τώρα πρέπει να δούμε πώς εξειδικεύονται αυτές οι αποφάσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα θα έχω τη δυνατότητα να κάνουμε σήμερα μια ε, ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων για τα δύο ε, χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναπτυξική συνεργασία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Συνεργασία για την Ανάπτυξη. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην στρατηγική μας, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη είναι κρίσιμη σημασία. Χρειάζεται να εμπεδώσουμε αυτή την ε, συνεργασία, να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί η καιρή είναι δύσκολη, το βλέπουμε τους τελευταίους ε, μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, πόσο έχουν δοκιμαστεί και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές αξίες από την μετανάστευση, από από τις συγκρούσεις, από τη μεσαλλοδοξία και την άνοδο του εξτρεμισμού που θέτουν σε κίνδυνο τις κοινωνίες μας και τις αξίες τους. Καθώς επίσης και τις ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει στην με την αναπτυξιακή συνεργασία να βοηθάει ανθρώπου στις πιο φτωχέ περιοχές του πλανήτη. Και αυτό συνεχίζει να το κάνει. Αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τους πόρους της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει την αφοσίωσή της στις ευρωπαϊκές αρχές. Και πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά να έχουμε μια τέτοια επικοδομητική προσέγγιση, να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα μακροπρόθεσμα προβλήματα, τις γενουσιουργές αιτίες της φτώχειας ή των προβλημάτων ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Μετά την δραματική αύξηση του αριθμού των μεταναστών και την προσφυγική κρίση δημιουργήθηκε το Ταμείο Εκτεκτής Ανάγκης για τους Πρόσφυγες που είναι ένα παράδειγμα που δείχνει με τον, οποίο, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει εργαλεία υφιστάμενα της, ε, της αναπτυξιακής συνεργασίας σε ευαίσθητες περιοχές του κόσμου όπως η Αφρική και να ενισχύσει τις προσπάθειες της ανταποκρινόμενη σε μια εκτακτή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια του 2014 περάσαμε μια μεταβατική περίοδο. Εκείνη την κατά τη διάρκεια του 2014 δεν είχαμε όλους τους πόρους στη διάθεσή μας για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ωστόσο συνεχίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες προγραμματισμού και καταλήξαμε τελικά στην Εστερική Συμφωνία που εγκαθίδρυσε το 11ο Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο για την Ανάπτυξη. Όμως τώρα μόλις έχουν, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση από την πλευρά των κρατών μελών, σιγά σιγά ε, ε ξεκινούν αυτά που από τη δικιά τους πλευρά πρέπει να κάνουν και περιμένουμε ότι θα είναι έτοιμα στο δεύτερο εξάμεινο του 2016. Κατά τη διάρκεια του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε ε, από τη δική της πλευρά πρωτοβουλία για να ενισχυθεί το, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δώσαμε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, εκφράζει την άποψή του να ε, γνωμοδοτεί επί των προγραμματικών ε, εγγράφων, των προγραμμάτων. Και γι' αυτόν τον λόγο επισκέπτομαι και κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων ε, μαζί σας κάθε χρόνο στην Επιτροπή σας. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι λειτουργεί αυτή η συνεργασία. τα τελευταία χρόνια θα σας δώσω ορισμένους αριθμούς. Στείλαμε 79 προσχέδια προγραμμάτων 71 ήταν ε, εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και 5 ήταν περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα, ενώ επίσης υπήρξαν και δύο ενδεικτικά προγράμματα που αφορούσαν περισσότερες ε, χώρες, περισσότερες της μίας χώρες, ε, το ένα για τις περιοχές του, Ανατολικού Τιμόρ και μετά για τις χώρες του ΑΚΕ. Παραμένουν επίση και κάποιε άλλε συζητήσει ακόμα να γίνουν για το ενδεικτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, για την Κεντρική Αφρική. Μετά από πρόσκληση τη ε, Κοινοβουλευτική σα Επιτροπή, επίση κάναμε συζητήσει και ανταλλαγή απόψεων για τα ε, ενδεικτικά προγράμματα ε, για το Κονγκό, για την Κάμπια, για το Λεσότο, για τη Λιβυρία, του Ζιμπάμπουε, καθώ επίση και για δύο περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα για την Κεντρική Αφρική και την Καραϊβική. Επίσης, ε, έγινε και μια γραπτή ανταλλαγή ε, απόψεων νομοδοτήσεων με την Επιτροπή σας για τρία εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, για επτά μάλλον ε, εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και τρία περιφερειακά. Τα εθνικά ήταν αυτά που αφορούσαν στην Αγγόλα, τον Βενίν, του νήσου Κομόρου, την Ερυθρέα, τον Μαλάουι, το Μαλί και την Μοζαμβίκη και τα περιφερειακά αφορούσαν την Κεντρική Αφρική, την Δυτική Αφρική, την Ανατολική Αφρική και τον ειδικό κενό. Συχνά τα θέματα που θέτει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι ε, τα ίδια. Ε, είναι κάποια που επανέρχονται. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ε, συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων. Είναι κάτι το οποίο τέθηκε και για τον Πενίν και για το Μαλί και τη Μοζαμβίκη και το Ζιμπάμβουε ε, και αλλού από την πλευρά μου δεν μπορώ παρά να τονίσω την σημασία που αποδίδουμε στην συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, επιτόπου, και των εθνικών κοινοβουλίων. Ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε μία από αυτές τις χώρες εταίρους. Πάντα κάνουμε μία ε, διαδικασία διαβούλευσης ε, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος και αυτή η διαδικασία διαβούλευσης ε, αποτυπώνεται και στα ενδεικτικά προγράμματα σε χώρες όπως για παράδειγμα η Μοζαμβίκη και το Ζιμπάμπουε, η διαβούλευση έγινε παράλληλα με διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για τον ρόλο που θα είχε η κοινωνία των πολιτών στην υλοποίηση του προγράμματος. Και δημιουργήθηκαν ε, κοινά εργαλεία για να παρακολουθείται η πρόοδο. Όμως η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών δεν σταματάει με το στρατηγικό προγραμματισμό πρέπει να συνεχίσετε και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Γιατί πιστεύουμε ότι τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται αποτελεσματικά μόνο όταν εφαρμόζονται από ε, τους τοπικούς φορείς. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ε, θεσμική κατάσταση στη χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, στο Μπενίν το Εθνικό Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά ε, στην επιλογή των τομέων εστίασης. Όταν υπάρχει μια κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια χώρα την οποία αφορά το ενδεικτικό πρόγραμμα, πάντα εμπλέκεται. Όσον αφορά τώρα τα περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή ε, και των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, υπερεθνικών φορέων, περιφερειακών υπερεθνικών φορέων. Ανάλογα βέβαια και με την αντολία αυτών των οργανισμών. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πολλέ φορέ από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξη είναι το ζήτημα τη χρηστή διακυβέρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη καταπολέμηση τη διαφθορά. Ιδιαίτερα για τι χώρε τη Αγκόλα, τη Μοζαβίκη, του Ζιμπάμπουε, του Μαλάουι, τη Κεντρική Αφρική και τη περιοχή τη Δυτική Αφρική. Ε, πράγματι πρέπει να ακολουθούμε μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό φάνηκε στα ε, ενδεικτικά προγράμματα για το Μαλάουι και για τη Δυτική Αφρική. λαμβάνουμε υπόψη προβλήματα διαφθοράς ή κακή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στον τρόπο με τον οποίο τελικά αποστέλνουμε τα χρήματα. Ε, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Αγκόλα, επιλέξαμε να γίνει χρηματοδότηση επί τη βάση project εξαιτίας αυτού του λόγου. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται ε, είναι τα, τα η σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις μας, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες αυτές. Κάθε φορά θα πρέπει να αξιολογούμε ποιο είναι το κόστος της μη παρέμβασης. Εάν δηλαδή έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προκαλέσει αλλαγές και αν πρέπει να κινητοποιηθεί και να το κάνει αυτό γρήγορα, ε, επιγόντως, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Μοζαμβίκης. Επίσης σας επισημαίνω ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται και με τη συνεργασία των δύο χρηματοδοτικών μέσων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη και του Ταμείου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα τη ζητήματα του φύλου ε, που ετέθησαν για το Λεσότο, για τη Μοζαμβίκη και για την Κεντρική Αφρική. Θα γνωρίζετε το ζήτημα της ε, ενδυνάμωση τη ισότητας των δύο φύλων, το gender mainstreaming, είναι κάτι το οποίο τίθεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, σε όλα τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα συμπεριλαμβάνουμε και μια ανάλυση της ισότητα των δύο φύλων, gender analysis. Ε, στην περίπτωση της Μοζαμβίκης έχουμε καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα ζητηθεί να εφαρμοστεί από το Υπουργείο για τις γυναίκες, τα παιδιά και την κοινωνική πρόνοια με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε επίσης να έχουμε δείκτες που να μας δείχνουν την ισότητα των δύο φύλων, κατά πόσον αυτή γίνεται σεβαστή, διατομεακούς και πιο συγκεκριμένους. πιο συγκεκριμένου δείκτες που να αφορούν συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, υποστηρίζονται οι γυναίκες, οι θεσμικές αλλαγέ που έχουν γίνει, εκπαίδευση ε, μεών κτλ. Στο Λεσότο, το ίδιο. Έγινε μια μελέτη για την ε, ισότητα των δύο φύλων που ενσωματώθηκε στο σχετικό σχέδιο. Γνωρίζετε ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές μου και της Επιτροπής. Η έννοια του gender mainstreaming και της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων έχει γίνει πλέον υποχρεωτική από τον Οκτώβριο του 2015. Αλλά αυτό για να εφαρμοστεί στην πράξη πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες στο επίπεδο το θεσμικό, αλλά επίσης και σε πρακτικό επίπεδο χρειαζόμαστε πόρους και ανθρώπινους και οικονομικούς η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει θέσει επίση το ζήτημα τη κοινωνική προστασία, τη κοινωνική πρόνοια για τι χώρε του Λεσότου, του Μπενίν, του Μαλή, τη Κεντρική Αφρική και τη Δυτική Αφρική για τα σχετικά ε, περιφερειακά προγράμματα. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω στην, στην ατζέντα για την αλλαγή. Ε, ε έχουν οριστεί κάποιες αρχές με βάση την ε, επικουρικότητα και τη συμπληρωματικότητα που θα πρέπει να έχουν τα προγράμματά μας σε σχέση με τις εθνικές πρωτοβουλίες. Και αυτό γίνεται σεβαστό σε όλα τα προγράμματα που αφορούν την Κεντρική Αφρική. Στη Δυτική Αφρική υποστηρίζουμε δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων και για την αντιμετώπιση των καταστάσεων μετά από μια κρίση, ε, ιδίως στα ζητήματα της ε, υγείας. το Λεσότο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μία από τις επιτυχίες μας ε, κατά τη διάρκεια του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους κατά το 11ο EDF. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ε, κυβέρνησης να βοηθήσει τις πιο φτωχές ε, κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα τους Μπασότο. Στην περίπτωση του Μαλή και στην περίπτωση του Μπενίν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επεμβαίνει άμεσα στην διάρθρωση του συστήματος υγείας αυτές τις χώρες με βάση την κατανομή εργασίας που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στη χώρα και στους διεθνείς δωρητές. Ένα άλλο θέμα που έχει τεθεί είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των παρεμβάσεών μας, ιδιαίτερα για το ζήτημα του Λεσότο. Ε, ιδιαίτερα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μεγάλα έργα σας διαβεβαιώνω ότι πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας το ζήτημα αυτό, ε, σε οποιαδήποτε παρέμβασή μας, είτε το έργο είναι μεγάλο είτε είναι μικρό, ιδιαίτερα ε, στην διαχείριση των υδάτων. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους δωρητές, θέμα που έχει τεθεί για την Αγκόλα, την Κάμπε, την Ερυθρέα και το Μαλάουι. Γνωρίζουμε ότι εδώ συνεργαζόμαστε, ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τι χώρε αυτέ σε ένα δύσκολο διεθνέ περιβάλλον. Επιμένω, προσπαθούμε να κρατήσουμε το διάλογο μαζί του ανοιχτό. Το να επιλέξουμε να μην παρέμβουμε θα είχε δραματικέ συνέπειες για τον πληθυσμό άμεσα, αλλά επίση και μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα για την σε, σταθερότητα στις περιοχές αυτές. Στην περίπτωση του Μαλάουι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι διεθνείς δωρητές και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη συμφωνήσει σε πιο πρακτικές ε, παρεμβάσεις που θα αφορούν κυρίως την λογοδοσία στο εθνικό επίπεδο, τη ε, διατροφή, την, την, την αντιμετώπιση των κρίσεων και την κοινωνική πρόνοια. Θα έρθω τώρα... Τρία ακόμα συγκεκριμένα στοιχεία για τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα των Κομόρο, καταρχάς. Αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υλοποίησης και χρειάζονται επαρκή ταυτοποίηση και σύνταξη και συμπλήρωση και αυτά τρέχουν. Για την Ερυθρέα. Η Κομισιόν παρότι μοιράζεται τις ανησυχίες που έχει και το Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση αυτή θεωρεί ότι η δέσμευση δημιουργεί τις δυνατότητες για να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για αλλαγές και πρόοδο συνολικά και να επιμείνουμε στην σημασία της αιμονής στα διεθνή πρότυπα και στη συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τον πληθυσμό και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις συνδίκες διαβίωσής του, όπως και τις συνδίκες σταθερότητας της χώρας και της ε, περιφέρειας. Τα χρήματα αυτά θα πάνε ή στο λαό της Ερυθρέας και όχι στην κεντρική κυβέρνηση. Ούτε στον τομέα της ενέργειας, ούτε στον τομέα της διακυβέρνησης και η Κομισιόν αυτά θα τα επιτηρήσει αυστηρά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φανεί ότι η ευρωπαϊκή πόρη, η βοήθεια, είναι βοήθεια προς το καθεστώς. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα κοινοβουλευτικά σχόλια ε, στα πλαίσια της 11 της CDF, θα μας καθοδηγήσουν και κάποιες αρχές προς τι οποίε έχουν συμφωνήσει τα μέλη της Επιτροπής EDF, μεταξύ των οποίων η αποτελεσματική υλοποίηση της περιοδικής αναθεώρησης των ΗΠΑ, που έχει αποδεχθεί η Ερυθρέα, και απτή πρόοδο στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη μεταρρύθμιση της στρατιωτική εθνικής θητεία. Το δε τρίτο θέμα αναφέρεται στα μέσα ανάπτυξης και συνεργασίας. Εδώ έχουμε διαφορετικές νομικές βάσεις. Πέραν του EDF επί του οποίου έχουμε συμφωνήσει ε, για ένα στρατηγικό διάλογο και υποτένει αυτή θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΔΕΒΕ και τα μέλη της για την συμμετοχή της στο στρατηγικό διάλογο DCI. Έχουμε όλοι επιφαληθεί από την πολύ καλή αυτή δουλειά διότι έχει ανοίξει θετικές οδούς πρόοδου για τον προγραμματισμό. Και προσμένω με ενδιαφέρον και την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις περαιτέρω συμφωνίες στρατηγικού διαλόγου που θα έχουμε μαζί σας, προτού γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική επανεξέταση του εγγράφου. Στο μεταξύ, και μετά τη συμπλήρωση του στρατηγικού διαλόγου και τη υιοθέτηση των εφάσεων της Κομισιόν για, για τον πολιετή προγραμματισμό, Βρισκόμαστε τώρα στη φάση της υλοποίησης. Και με χαρά θα συνεχίσουμε τον τακτικό αυτό διάλογο μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων και για να ολοκληρώσω να επαναλάβω τις θερμές ευχαριστίες μου για τις πολύ καλές ερωτήσεις και την πολύ καλή εξέταση διαθεσμικά που παρήχατε. Πρόκειται για μια αμοιβαία διαδικασία συλλογής εμπειρίας και μάθησης. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε τον Επιτροπό που υπήρξε τόσο συγκεκριμένος για τις απαντήσεις επί των, από, επί των συγκεκριμένων επιστολών που είχε λάβει από τα μέλη. Εδώ έχουμε συντονιστές από τις διάφορες επιτροπές και έχουμε και κάποιους από τους προέδρους των ε, ομάδων εργασίας όπως ζητώ συγγνώμη γιατί μπορώ να τον κατάλογο της Κεντρικής Ασίας, των παγκοσμίων προκλήσεων Αφ... Αφρικής και Ινδικού Ωκεανού όπως και της ε, Νότιας Ασίας, ανθρωπιστικής βοήθειας και εθελοντών. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ΕΛΚ. που είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα βέβαια στο Κοινοβούλιο. Μετά θα πάμε στο συσιοσιαστική ομάδα. Θα, πάμε, θα πάρουμε τους τρεις πρώτους και μετά θα δούμε πόσες ερωτήσεις θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα πάρουμε τις πρώτες τρεις και μετά άλλη μια ομάδα τριών ερωτήσεων ώστε να δώσουμε και την ευκαιρία στον Επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους της ε, από από το Κοινοβούλιο, την ε, Κομισιόν και να επαναλάβω αυτό που είπε ο πρόεδρος από την αρχή, ή πρόεδρος, στο συγγνώμη, από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Να ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε το τελευταίο χρόνο που κυρίως επικεντρώθηκε στη νέα δέσμη στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα θέλαμε μάλλον αυτά εναρμονίστηκαν και ενεκρίθησαν το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια και φέτος είμαστε βέβαιοι ότι η εστίαση θα είναι επί της υλοποίησης. Η Κομισιόν το έχει τονίσει αυτό αρκετές φορές ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουμε με αένα ψηφίσματα αλλά να εστιαστούμε περισσότερο ή στην παρακολούθηση, την επιτήρηση των ε, ήδη υφισταμένων προγραμμάτων και στην υλοποίησή τους. Η Επιτροπή αυτή πάντοτε παρήχε στήριξη για μια πιο ισχυρή, πιο συνεκτική πολιτική ανάπτυξης και θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή υπογραμμίζοντας ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια συνεκτική και σταθερή και αποφασιστική πολιτική, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς που διατρέχουμε. Παρότι βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Η συνεργασία βεβαίως μεταξύ της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είχε ένα πεδίο δυνητικής βελτίωσης και θα αναφερθώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσατε. Έχουμε και κάποια τεχνικά ζητήματα, όπως οι προθεσμίες για την υποβολή εγγράφων από πλευράς κομισιών προς την Επιτροπή. Θεωρώ ότι αυτές οι προθεσμίες είναι αρκετά στενές και ίσως εδώ θα μπορούσαμε κάπως να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γιατί πέρα από την τεχνική του διάσταση αυτό θα επιτρέψει τα μέλη να πραγματοποιήσουν την ουσιαστική επιτήρηση που ζητεί και η Κομισιόν. Και σε σχέση με την επιτήρηση αυτή και στο πλαίσιο των πολιετών προγραμμάτων πάντοτε υπάρχει χώρος βελτίωσης, περιθώριο βελτίωσης. Ωστόσο η Κομισιόν δεν απήντησε στην πρόσκληση των ομάδων εργασίας της Επιτροπής αυτής. Πιστεύουμε βεβαίως ότι η ίδια νομική βάση που έχουμε για τα πολιετή προγράμματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα ετήσια προγράμματα δράσεως τα οποία όπως είδαμε και στην περίπτωση της Ερυθρέας στην οποία αναφερθήκατε εκτενώς θα είναι ακριβώς στο επίκεντρο της εστίασης της δουλειάς, της κοινή δουλειάς, Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν θα πρέπει να προσέρχονται στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας. Υποβάλλονται και τις πληροφορίες σχετικά με διάφορα προγράμματα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω διαθέσιμου εγώ, υπήρξαν αιτήματα και από την υπηρεσία εξωτερική δράσεω για ενημέρωση και θεωρώ πως θα έπρεπε συνολικά να απαντάει η Κομισιόν πιο έγκαιρα σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και αιτήματα. Σε σχέση με την περίπτωση τώρα της ε, συγκεκριμένα της Ερυδρέας και τα συμπράσματα του Κοινοβουλίου μπορούμε να συζητήσουμε τον περιεχόμενο. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες ε, πτυχές. Τα κράτη-μέλη δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς, επαρκώς λέω, σχετικά με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άρα τα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε κράτη-μέλη προκειμένου τα κράτη-μέλη να είναι απολύτως ενημερωμένα και επί τη βάση της ενημερώσεω αυτή να μπορούν και εκείνα να φτάνουν σε χρήσιμα και ενημερωμένα συμπεράσματα. Ή στην περίπτωση της Ερθρέας, εξ όσων εγώ γνωρίζω, δεν συνέβη έτσι. Και τα κράτη-μέλη είτε είχαν λανθασμένη πληροφόρηση, είτε δεν είχαν καθόλου πληροφόρηση σχετικά με την αντίρρηση του Ευρωκοινοβουλίου προς την έγκριση του εγγράφου αυτού. Είχα σημειώσει και άλλα δύο θέματα, αλλά θα αναφερθώ σε ένα. Είπατε ότι το 2016 θα είναι το έτος της έναρξης του νέου διαλόγου για την συνένεση επί της ανάπτυξης. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε πώς αυτό θα διαρθωθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Αντίκη Γερέρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, εκτεταμένη αυτή παρέμβαση και τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε σχετικά με τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα και το πώς αυτά λειτουργούν. Εγώ συμφωνώ με αυτό που ανέφερε ο Ντάβορ ότι το 2016 θα πρέπει να είναι το έτος της εφαρμογής, της υλοποίησης πολλών από τις γραμμές που ανοίξαμε κατά τη διάρκεια του έτους 15, το οποίο έτος είναι ανεπανάληπτο, θα λέγει κανείς, υπό την έννοια της ε, έναρξης, της ε, δημιουργίας διαφόρων πολιτικών ανάπτυξης, συμφωνίες που υπεγράφησαν, δεσμεύσεις που ανελήφθησαν, η σύνοδος κορυφής ανθρωπιστικών θεμάτων που θα λάβει η χώρα το Μάιο ή στην ε, Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει το 2015 επεξεργαστήκαμε την βασική δομή και αρχιτεκτονική της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη για την ερχόμενη περίοδο διαφόρων ετών. Και τώρα θα πρέπει αυτά να τα εφαρμόσουμε και θα πρέπει η Κομισιόν και η Επιτροπή Ανάπτυξης να συνεργαστούμε προς την εφαρμογή και την υλοποίηση των ζητημάτων αυτών. Δευτερευόντως θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα επί του είδους της εργασίας που καλούμαστε να αναλάβουμε ε, στα πλαίσια των καθηκόντων αυτής της παρακολούθησης που διενεργούμε σήμερα. Αυτή η παρακαλούθηση, αυτή η επιτήρηση είναι μία από τις βασικότερες λειτουργίες του κοινοβουλευτισμού γενικά θα έλεγα και είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα διήβρινε την νομοθετική του αν θέλετε αρμοδιότητα αλλά αυτό θα πρέπει παράλληλα να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι περισσότερο αναγνωρίσιμο ως προς τις διαδικασίες αυτής παρακολούθησης και ως προς τις τακτικές του επαφές με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και άλλους θεσμούς. Εν πάση περιπτώσει ανταλλάγουμε πληροφορίες, καλώς το κάνουμε αυτό και η Κομισιόν οπωσδήποτε έχει την ευκαιρία να καταλαβαίνει τις τάσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου γενικά. Το Ραουντάβορ αναφέρθηκε σε μια σειρά από προβλήματα. Δεν θα επιμείνω εγώ περισσότερο σε αυτά που εκείνος ανέπτυξε. Όμως έχουμε εκείνο το ζήτημα πράγματι των πολύ στενών προθεσμιών που έχουν τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσουν τα, τις προτάσεις και τα έγγραφα προγραμμάτων των ε, προαιρετών ε, ενεξελίξη προγραμμάτων που υποβάλλει η Κομισιόν. Τώρα ε, αυτά τα στοιχεία ενδεχομένω για την Κομισιόν να μην είναι απολύτω εμφανή και πρώτη ε, θέλετε πρώτου επίγοντος αλλά είναι οπωσδήποτε εμφανή για εμάς. Δεν είμαστε αναγκαστικά όλες τις ημέρες της εβδομάδος σε συνάντηση και το οποίο σημαίνει ότι επί τη βάση του χρονοδιαγράμματος που έχουμε εγκρίνει στην προηγούμενη Ολομέλεια και μιλώ για το πρόγραμμα το κοινοβουλευτικό για το 2016 το ετήσιο και αν συμβούν τα ίδια με αυτά που συνέβησαν πέρυσι θα έχουμε 9 εβδομάδες ε, κοινοβουλευτικής ε, πολιτικό Δραστηριότητα με επισκέψει στι πρωτεύουσε, στι χώρε κτλ. κτλ. Εμάστε στι εκλογικέ περιφέρειε. Α μην επαναλάβουμε την συζήτηση που είχε ήδη λάβει χώρα. Αν τώρα αποκλείσουμε τι εβδομάδε αυτέ, τι οποίε πρέπει να αφιερωνόμαστε στι χώρε μα. Εάν εξαιρέσουμε τι θερινέ, περιόδους, τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, και κάποιες άλλες περιόδους εν πάση μέσα στο έτος εάν λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, οι προθεσμίες και τα περιθώρια τα χρονικά που έχουμε είναι πάρα πολύ περιορισμένα προκειμένου να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε δουλειά αυτής εδώ της σημασίας. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που να πούμε ότι τα έγγραφα που αποστέλει η Κομισιόν τα αποστέλει είτε με καθυστέρηση είτε την Πέμπτη πριν από ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Τώρα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες προθεσμίε επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει και προβλέπουν οι κανόνε σε πάση περιπτώσει. Και ότι δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τους κανόνες. Όμω, αρκετά μέλη τη αίθουσα αυτή θα ήταν πολύ ικανοποιημένα εάν λαμβάναμε υπόψη μας εντό των προθεσμιών αυτών τι αποτελεσματικέ, τι διαθέσιμε ημέρε κοινοβουλευτική εργασία δεδομένα των υποχρεώσεών μας. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιούμε περισσότερο την γραπτή διαδικασία η οποία περιορίζει το χρόνο εντός του οποίου πρέπει να απαντούμε προς την Κομισιόν. Και να συμφωνήσω επίσης με τον Ντάβορ σχετικά με την παρουσία της Κομισιόν των εκπροσώπων της Κομισιόν ή στις ομάδες εργασίας της Επιτροπής όταν κοιτάζουν τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι Τώρα μπορεί να μπερδευτεί κανείς και στα ισπανικά και σε άλλες γλώσσες μεταξύ της Επιτροπής, της Κομίσιον, της Κομισιόν και τα ρέστα. Εν πάση περιπτώσει η Κομισιόν έχει πολλά να κερδίσει παρακολουθώντας τις εργασίες των ομάδων εργασίας μας. Θα ήταν πολύ επικοδομητική η παρουσία της. Και όχι μόνο θα ήταν ένα στοιχείο πρόσθετης ενημέρωσης για την Εκτελεστική Επιτροπή, λέει ο μιλητής, για την Κομισιόν, αλλά θα αναπτύσσαμε ένα, μια ατμόσφαιρα συνεργασίας, ένα κλίμα καλύτερης συνεργασίας και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα είχαμε κάποιες αντιρρήσεις ή κάποιες τροπολογίες που υποβάλλονται κτλ. Εφόσον δηλαδή θα υπήρχε αυτός ο άμεσος διάλογος και αυτή η άμεση συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν και της Επιτροπής μας. Τώρα, συμφωνήσαμε ακόμα δεν έχουμε εγκρίνει επισήμω, το νέο, τη νέα συμφωνία διαθεσμικής συνεργασίας και εκεί υπάρχει μια σειρά από στοιχεία σχετικά με τη διαφάνεια, την συνεργασία, τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά κτλ. Δεν θα προσθέσω τίποτα επί της Ερυθρέας γιατί έχω την εντύπωση ότι ήδη συζητήθηκε αυτό σε διάφορες συναντήσει της ε, Κομισιόν και θυμάμαι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ε, που είχαν αναφερθεί οι συνάδελφοι άμεσα και ευθέως στο θέμα αυτό. Απλώς λοιπόν θα πω ότι συμφωνώ με την ε, θέση αρχής που εξέφρασε ο κύριος Νίμισα Όταν υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις ή συγκρούσεις, τότε δεν διεξάγεται καλά η συνεργασία. Το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε τη συνεργασία μας αυτή, προκειμένου να πείσουμε την άλλη πλευρά να υιοθετήσει, αν θέλετε, αποφάσεις που δεν θα υιοθετούσε αν δεν ήταν υποπίεση. Αλλά βεβαίως αυτή η πίεση πρέπει να ασκείται με όρια που θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση όταν έχουμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Δηλαδή, συνεργασία βεβαίω, αλλά θα πρέπει επίσης να είναι σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Και κάτι ακόμα σχετικά με αυτήν τη νέα συμφωνία διαθεσιμική συνεργασίας θα πρέπει να περιοριστεί η το ελάχιστο η εμπιστευτικότητα των εγγράφων ή αν θέλετε η υπερβολική χρήση της εμπιστευτικότητα αυτής διότι αυτό μειώνει την δυνατότητα αυτή τη σωστή και αποτελεσματική παρακολούθηση πρέπει να διεξάγει το Κοινοβούλιο. Εμεί λοιπόν κύριε Επιτρόπε βλέπουμε θετικό μάτι την συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής με την ε, Κομισιόν. Ήθελα απλώ να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που όλες οι ομάδες νομίζω συμφωνούμε ότι μπορούν να βελτιωθούν και θα βελτιώσουν και τη συνεργασία των δύο πλευρών. Έχω βέβαια μακρό κατάλογο ομιλητών, τον Σαρλ ε, Γκέρενς πρώτα. για, για σας ε, της Βουλής των Κοινοτήτων λέω ότι είναι από του φιλελευθέρου. Ε, κανείς δεν είναι τέλειο τέλειος λέει ο κ. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω με την σειρά μου τους εκπροσώπου ε, τη Βουλή των Κοινοτήτων απέναντι στο έργο στην αναπτυξιακή βοήθεια που κάνει το Ενωμένο Βασίλειο μένουμε πραγματικά έκθαμβοι είστε εκπρόσωποι μια από τις σπάνιες εκείνες χώρες που τήρησαν τα υπεσχημένα και που υλοποιεί τις υποσχέσεις της και λέει και τα όσα έπραξε. Επαναλαμβάνω ότι σας θαυμάζουμε για, την, ε, για το κατόρθωμα σας αυτό και μάλιστα σε μια περίοδο και δημοσιονομικής λιτότητας. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. καλώς έκανε να εισαγάγει τη συζήτηση ο Επίτροπος βάζοντας επιτάπητος σε διάφορα θέματα που έχουν ενδιαφέρον για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί το κοινοβουλίο μας. Έχουμε σε κάποιες μεταβλητές που θα έχουν επίπτωση στο κλίμα μέσα στο οποίο θα εργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. Και πρώτα αυτός ο πολλαπλασιασμός των Trust Fund στην Μάλτα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δώσει 3,5 δισεκατομμύρια στην Αφρική στα πλαίσια του Trust Fund για την Αφρική. Η Κομισιόν κινητοποιεί τους πόρους τους οποίους αντλεί από το ε, από θεματικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως εκεί δεν έχω κάνει καμία αντίρρηση και θα προσφέρει επίσης οι χώρες, θα προσφέρουν οι χώρες μέλη 1,8 δις όμως δεν προσφέρουν τίποτα, 5% το πολύ. Εδώ και μήνες μένουν σε αυτή την ε, πάρα πολύ μετριοπαθή συνεισφορά και δεν φαίνεται πουθενά κάποιο φως ελπίδας ότι θα αυξήσουν την συνεισφορά τους. Τι θα κάνετε 3,5 δισεκατομμύρια εάν δεν χρηματοδοτηθούν, θα τα μειώσετε στο μισό το Trust Fund που κρίνει αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει στην ανταπόκριση των δυσχεριών που αντιμετωπίζει η Αφρική. Θα τα μειώσετε τα χρήματα αυτά ή θα προσπαθήσετε να βρείτε το εναπομένον 1,8 δις από κάποια άλλα συρτάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο, δεύτερη μεταβλητή, το χρέος της Αφρικής. Θεωρούσαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω το πρόβλημα. Όμως τώρα διαπιστώνουμε και το επιβεβαιώνουν εμπειρογνώμονες ότι το χρέος βρίσκεται ξανά σε αύξηση στην Αφρική. Πέραν μάλιστα και του ευρωπαϊκού ή μάλλον λιγότερο από το ευρωπαϊκό όριο, λιγότερο από το ευρωπαϊκό όριο, αλλά σε ορισμένα σημεία έχει φτάσει και σε ανισχυτικό σημείο. Και αυτό λοιπόν θα έχει επίπτωση και στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως. Τρίτο σχόλιο, ε, ή μάλλον μια αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως και τη νέα σχέση με τις χώρες Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού. ΑΚΕ. Στα πλαίσια μιας υγιούς ε, προσπάθειας προγραμματισμού θα χρειαστεί να έχουμε ξεκάθαρες ιδέες ήδη από τώρα σχετικά με το τι θα συμβεί μετά το 2020. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται να δεσμευτεί ένα μέρος των δαπανών που δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα παρά μόνο στο μέτρο όπου θα είναι εξασφαλισμένη μια συνέχεια μετά το 2020. Ε, τέταρτη μεταβλητή. Ποια θα είναι η επίπτωση των ε, εμπορικών συμφωνιών, οικονομικών συμφωνιών στις δυνατότητες επενδύσεων στις αφρικανικές χώρες. Ε, επενδύσεις είτε σε βάρος των κρατών είτε σε βάρος ε, με χρηματοδότηση των ταμείων. <clears throat> Πώς κρίνεται την επίπτωση αυτή. Πέμπτο σχόλιο. το Παναφρικανικό πρόγραμμα πώς διαρθρώνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ε, αφρικανικές χώρες των ΑΚΕ. Αν θυμούμε καλά, πρόκειται για ένα δισεκατομμύριο ευρώ για το Παναφρικανικό σχέδιο, για το Παναφρικανικό πρόγραμμα, για μία περίοδο 7 ετών. Η ίδια επιτροπή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα αυτό θα είναι, αλλά πρόκειται για διαφορετικό εργαλείο που εμπίπτει στο DCI. Χρηματοδοτείται λοιπόν από το DCI. Α, αυτές είναι οι ανησυχίες που με διακατέχουν. Εκφράζω και πάλι την επιθυμία μας, παρουσία και των Βρετανών συναδέλφων μας, να δούμε τους υπουργούς συνεργασίας για την ανάπτυξη ή και των οικονομικών να προσέλθουν εδώ ενώπιον της Επιτροπής μας όπως γίνεται και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να αποδώσουν λόγο για τις δεσμεύσεις τους, τις οποίες έχουν αναλάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη και που νομίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη λέει ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε ακριβώς ό,τι έχουμε υποσχεθεί και θα τηρήσουμε το λόγο μας. Θα τιμήσουμε την υπογραφή μας. Αυτό θα έπρεπε να είναι το μοναδικό σύνθημα, ο μοναδικός τίτλος του προγράμματος αυτού διότι από το 2005 μας λένε παραμύθια τα οποία δεν πιστεύουμε πλέον. Χρηματοδοτήσεις για την Τουρκία, για παράδειγμα. Βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο της χρηματοδότησης από τις χώρες μέλη. Μόλις πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα στην ρίζα του, βλέπουμε αυτήν την αποστασιοποίηση. Είναι δυνατόν να μας πάρουν στα σοβαρά όταν λέμε τα ίδια πράγματα αυτά. Με ναι, τη συνεργασία των κρατομερών και του Κοινοβουλίου πρέπει να μετακινηθούν οι θέσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι φτάνουμε σε κάποια όρια των δρασεών μας. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τον τόνο, θα πρέπει να αναζητήσουμε μια πιο αποτελεσματική μέθοδο, μεθοδολογία αν θέλετε, ώστε να εμφανιστούμε και πιο αξιόπιστοι στα όματα των συνομιλητών μας, οι οποίοι κρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι και αυτό αποτελεί μέρος της συζητήσεως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία ε, εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτό. Νίρς Ντέβα από την Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Εμένα με διακατέχει το αίσθημα ότι τα έχω ξαναδεί και τα ξανακούσει αυτά τα πράγματα. Δέκα χρόνια είμαι εδώ και μου φαίνεται ότι ξαναλέμε τα ίδια. Έχουμε όλα τα εργαλεία επιτάπητος, μιλούμε για προγράμματα, για χρηματοδοτήσεις, πώς να παρακολουθούμε, πώς ε, θα εξευρεθούν οι πόροι, διάφορα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και συνεχίζουμε με την ίδια τακτική. Έρχεται ο Επίτροπος και μας τα λέει ωραία και με γλαφυρό τρόπο και όπως έκανε μόλις τώρα ο Επιτρόπος Μίμητσα και εμείς λέμε λίγα από εδώ, λίγα από εκεί και συνεχίζουμε. Έχω την έκθεση εδώ της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Πραγματική καταστροφή. Λέει ότι υπάρχουν επιτόπου χρήματα της Ένωσης που δεν φτάνουν στο στόχο τους. Ότι υπάρχουν αντιπροσωπείες που δεν αποδίδουν στο έργο τους ότι σπαταλώνται χρήματα σε τεράστιες ποσότητες. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όλες οι αντιπροσωπείες στα τέλη του 2014 είχαν ποσά 20,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αδιάθετα. Τα χρήματα για να διατεθούν αυτά τα αδιάθετα χρήματα θα χρειάζονταν λοιπόν 3,8 χρόνια. Με το ρυθμό αυτό όμως θα χρειαστούν οι αντιπροσωπείες 27 χρόνια για να ρευστοποιήσουν τους πόρους που διαθέτουν. Όπως είπα 28 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσμπεκιστάν, 16 χρόνια για παράδειγμα. Αζερβαϊτζάν. Για ποιο λόγο δίνουμε χρήματα στο Αζερβαϊτζάν, αλλά να που δίνουμε χρήματα στο Αζερβαϊτζάν. Άλλα, πάλι 16 χρόνια. 123 εκατομμύρια. Από τις πιο πλούσιες σε του κόσμου τα Αζερβαϊτζάν, έτσι. Και άλλου 14 χρόνια. ...2.598 ε, project έργα τα οποία υποειλοποιούνται άλλα 105 έργα, πάλι τάξιος πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, των οποίων η εκτέλεση καθυστερεί. Καθυστερεί η δαπάνηση κάθε δεύτερου ευρώ. Δηλαδή από τα δύο ευρώ το ένα καθυστερεί να δαπανηθεί και δεν φτάνει στον αρχικό στόχο του. Μιλάμε για κόκκινες γραμμές. Α, ή κόκκινα φώτα και ε, έχουμε το κάθε τρίτο ευρώ δεν έχει την σχεδιαζόμενη επίπτωση. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 68 ε, έργα καθυστερούν και δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ τους αρχικούς τους στόχους. Κύριε Πίτροπε, εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ αν με βάρενε ένα τέτοιο έγγραφο να ε, βαθμολογεί την απόδοσή μου. Όταν βαθμολογούμε τις διάφορες αντιπροσωπείες, αν τα πάνε καλά ή λιγότερο καλά, πολλές από τις αντιπροσωπείες μας, δυστυχώς και της χώρας όπου γεννήθηκα, τα πάνε χειρότερα. Έχουμε βάλει τώρα επιτροπές ε, παρακολούθησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα, αλλά βρισκόμαστε σε κρίση, κύριε Επίτροπε πρέπει να επανείδουμε, να επανεξετάσουμε κάθε ένα από τα, τα έργα αυτά. Πρέπει να στείλουμε κόσμο να δούμε πού πάνε τα λεφτά αυτά ή μάλλον πού δεν πάνε. Και αν δεν πάνε τα λεφτά αυτά, το γιατί, γιατί πράγμα μιλούμε. Όσο τα λεφτά δεν πάνε στο σκοπό του, πεθαίνουν άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, είτε από την πείνα, είτε από την λειψιδρία, είτε από τι ασθένειε. νομίζω πρέπει εδώ να ανάψουμε το κόκκινο φως και να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να αναλάβουμε επιτέλους δράση. Η πρόεδρος Άβαν, ευχαριστώ. Για την έκθεση που αναφέρατε, δεν είναι έκθεση της Επιτροπής Έλεγχου Προϋπολογισμού, είναι σημείωμα το οποίο έχει συντάξει γραφείο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολισμού και το διάβασα εγώ στον τύπο, στην εφημερίδα. Δεν ήρθε ο πρόεδρος της Κοκομπή να μου τα πει αυτά τα πράγματα. Αν υπάρχουν προβλήματα με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια και γνωρίζει κάποιος και συντάσσει εγγραφών να έρθει να μου τα πει. Όχι να πάει να τα πει στους δημοσιογράφους. Και την Πέμπτη όταν συναντήθηκε στο Στρασβούργο η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού Δεν ετέθη το θέμα αυτό ε, εν ώψη και της ε, Πρόεδρου. Άρα δεν είναι επίσημο έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Εάν υπάρχουν θέματα, τα θέματα αυτά να συζητηθούν εδώ, να τεθούν από την ε, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, να προσέλθει εδώ σε μας και να τα συζητήσει μαζί μας. Είναι περίεργο που συναντάται ολόκληρη Επιτροπή πέμπτη πρωί και δεν τίθεται το θέμα αυτό από την Πρόεδρο και, τη, και ενώπιον της είπα της εκπροσώπου την οποία την είχε εκεί παρούσα. Γνωρίζω την, πώς να το πω, τη μελέτη αυτή, τα γνωρίζω όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι άλλα είναι αυτά τα πράγματα και άλλος ο επίσημος τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά. Δεν βασίζονται τα στοιχεία αυτά στην έκβαση των έργων βασίζονται στο πρώτο έτος της έναρξης εφαρμογής τους. Πρώτος χρόνος, όταν οι πρέσβεις λένε έχουμε ένα πενταετές έργο ή πρόγραμμα, εδώ βρισκόμαστε, έχουμε προβλήματα εκεί, εκεί και εκεί. Βεβαίω και έχουμε προβλήματα με τη Συρία, με την Ιεμένη, ασφαλώς, ε. Ας κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν προβλήματα σε τέτοιες χώρες. Σοβαρή συζήτηση για σοβαρά θέματα. Νέρς, θα επανέλθουμε στο θέμα σας. Η κυρία Χαουτάρα. Ευχαριστώ, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Λίντα Μακάβαν που είναι η πρόεδρός μας. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ σοβαρό κοινοβουλευτικό έλεγχο και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε με τον κύριο Μίμητσα και καλώ ήρθατε κύριε Επιτροπή. Δεν χρειαζόμαστε όμω τέτοιου είδου σκανδαλώδη συμπεράσματα που ενθουσιάζουν τι εφημερίδε. Μιλούμε και για αποτυχίες όπως, σε χώρες όπως Βανουάτου ή τα νησιά Σολομόντος, τα οποία, τι να πω, εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης από τους τυφώνες. Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε ως συνήθως με την εφαρμογή προγραμμάτων σε τέτοιες χώρες. Βεβαίως και η Συρία, η Εμένη, γνωρίζω ότι είναι, γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι οι πιο έφραστες, αποτυχημένες χώρες στον κόσμο. Χρειάζεται χρόνος για να στήθουν στα πόδια τους έργα σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι διόλου χρήσιμο να τα μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι τέτοια πράγματα τα οποία δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα ούτε έρχονται μετά από συζητήσεις των αρμοδίων οργάνων. Είναι ντροπή πραγματικά που η Επιτροπή, μάλλον η Πρόεδρος της Επιτροπής Ενόχου Προπολογισμού δεν προέδρευσε καν στη σχετική συνάντηση. Και τώρα να έρθω σε αυτά που λέχθηκαν ω τώρα για την διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου που νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία έχει επιτέλους αναλάβει και χρειάζεται να αποδώσουμε καλά και καλύτερα από ό,τι έως τώρα. Πιστεύω ακόμη ότι η ουσία εδώ είναι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερους τρόπους να προβάλλουμε επιχειρήματα και να συζητούμε και να μαλώνουμε ακόμη για αμφιλεγόμενα θέματα. Το περίφημα παράδειγμα των, ε, ε, του προγράμματος εθνικών δικτών για την Ερυθρέα το κοινοβούλιο είπε να μην ανακατευτούμε με την Ερυθρέα. Είπε ότι χρειάζεται ένας πιο καλά ε, στοχευμένος τρόπος για να ασχοληθούμε. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως πάνω σε κάτι, κύριε Επιτροπέ. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην είναι καν παρούσα στις συναντήσεις των ε, ομάδων κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν είναι σωστό ε, εσεί να βράτε εμείς να ε, επικρίνουμε. Το άλλο είναι το, η εμπιστευτικότητα των εγγράφων που δεν εξυπηρετεί τον στόχο. Δηλαδή δεν επιτυγχάνονται έτσι αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Εγώ ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το ε, Συμβούλιο για θέματα Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως να εξετάσουν προσεκτικά αν, υπάρχουν καν, αν υπάρχει καν νομική βάση στην νομοθεσία μας για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εγγράφων. Γιατί να είναι εμπιστευτικά τα εγγράφα αυτά. Έχει κάποια σχέση με κρατική ασφάλεια ή με την αποφυγή βλάβης σε διεθνείς σχέσεις. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης, χωρών μελών της και των χωρών εταίρων. Έχω τώρα ορισμένε ερωτήσεις σχετικά με τα ειδικά ταμεία ιδίως αυτά που ανέφερε ο κ. Γκέρενς. Υπάρχει λόγος ανησυχίας σήμερα. Χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί για την αναπτυξιακή βοήθεια τώρα μπαίνουν στη μέση και τόσα άλλα συμφέροντα. Τελικώς απευθύνουμε κατηγορίες σημαίνει στους δε, ενώ το Κοινοβούλιο χρειάζεται την Κομισιόν και το αντίθετο. Και αυτό που χρειάζεται είναι να επιτευχθούν αποτελέσματα. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, υπάρχει επιχείρημα σήμερα που να πείθει ότι πρέπει να διευκρινίσουμε για ποιο λόγο αυτά τα ειδικά trust funds διατίθεται. Χρειάζεται να ανησυχούμε για το γεγονός ότι τα δημόσια χρήματα που δίνονται στην αναπτυξιακή βοήθεια κατά κάποιο τρόπο υφαρπάσονται από άλλους φορείς που έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως αυτά που προκαλούν τη μετανάστευση, το προσφυγικό κτλ. Αλλά χωρίς να προδώσουμε τις αξίες μας που συμπεριλαμβάνονται και στις αξίες του ΩΣΑ το γενικότερα τη διεθνού αναπτύξεω κτλ. Πάντω νομίζω κύριε Επιτροπέ, ότι χρειαζόμαστε όντω περισσότερο διάλογο. Και καλά κάνατε και ήρθατε εδώ να μα μιλήσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα σα πρότεινα να ακούσουμε όλε τι ερωτήσει από όλου του συναδέλφου και να δώσουμε στο τέλο το λόγο στον Επίτροπο, ο κύριο Φροντζούλητσα. Ιδιαίτερα δραστήριο στην ομάδα μα, ω γνωστό. Κύριο Φροντζούλητσα. Σα ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, Καλή χρονιά. Και ότι καλύτερο είναι το 2016. Ελπίζω να έχουμε και μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2016. Η ε, ομάδα εργασία μα ε, συναντήθηκε 7 φορέ. Καταλήξαμε σε συμπεράσματα για 12 θέματα, για εθνικά ε, ενδεικτικά προγράμματα και για περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα και τρία έγγραφα συμπερασμάτων για το DCI. Δεν θα επαναλάβω αυτό που ακούστηκαν για το ζήτημα της Ερυθρέας. Ήταν τελείως απογοητευτική ε, η κατάσταση. Ε, ήταν τελείως απογοητευτικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε την γνωμοδότησή μας. Μας χαροποιεί η συνεργασία. Είστε πάντα καλοδοχομένος, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ίδιο επίπεδο συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε καν ε, μας επιβεβαιώνουν ότι έλαβαν ε, ηλεκτρονικά τις ε, παρατηρήσεις μας. Ενώ ταυτόχρονα κάθε φορά που ε, ε, διαβάζουμε τα γραφά τους ε, διαπιστώνεται ότι καταγράφεται ότι λάβαμε σχόλια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποτέ δεν, διαπιστώ, δεν καταγράφεται ότι λάβαμε ε, αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ακριβώ αυτό το οποίο έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το EDF, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε και την ε, ε, συνεργασία μας μαζί σας γιατί είναι γνωστό ότι εσείς μεταβιβάζετε τις, διαβιβάζετε τις απόψεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, ποτέ δεν λάβαμε επισήμω ή ανεπισήμω μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρεκτός μια φορά για ένα περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα στο οποίο ε, οι υπηρεσίες δέχτηκαν να κάνουν μια τροποποίηση που είχαμε προτείνει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς διώκουμε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά και τις υπηρεσίες της, όχι μόνο με εσάς, και αυτό προκειμένου να αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά ταμεία και όλα τα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση των αξιών μας. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου. Αυτές πρέπει να προασπίζουμε με όποια χρηματοδότηση. Μιας και είναι παρόντες και οι συνάδελφοι από την Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, θα ήθελα να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η Βρετανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως γνωρίζετε ε, πολλές χώρες ε, ευεργετούνται από τα προγράμματα του EDF και εάν η Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπονομευτεί και η σημασία της στη διεθνή σκηνή. Βεβαίω θα είναι σημαντική, αλλά είναι πολύ σημαντικότερη σήμερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σημασία η παραμονή της Βρετανίας και για την, τα μέλη της Ένωσης και για την ίδια. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πράγματι θα κάνουμε μια σχετική συζήτηση, φαντάζομαι, με τους ε, προσώπους της Βουλής των Κοινοτήτων. Κυρία Γκραμπόσκα. Από την ομάδα εργασίας ε, για τη Μέση Ανατολή την Κεντρική Αφρική, την ΑΚΕ και άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον Επιτρόπο. Εκ μέρους της ομάδας εργασίας C θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για το έργο μας. Δυστυχώς αυτά που έχω να αναφέρω εγώ είναι πολύ παρόμοια με εκείνα που ανέφερε ο συνάδελφο Φροντζούλητσα από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Οκτώβριο του 2015. Εμείς εξετάσαμε πέντε προγραμματικά έγγραφα και καταλήξαμε σε γραπτά συμπεράσματα τα οποία ε, ενέκριναν οι συντονιστές της ε, Επιτροπής και ζητήσαμε περιπτέρω πληροφορία. Ζητήσαμε follow-up, περιπτέρω ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ασκήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών των προγραμματικών εγγράφων. Οι ανησυχίε μας ήταν κυρίως ότι δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε στην μείωση της φτώχειας ή την τήρηση των διεθνών προτύπων. Για παράδειγμα, είχαμε αντιρρήσει όσον αφορά την στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πρόγραμμα που αφορά τι χώρε ΑΚΕ Εδώ τέθη θέμα χρηματοδότησης. Μια άλλη ανησυχία της ομάδας εργασίας μας είναι ότι δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση ειρηνευτικών προσπαθειών στην Αφρική. Θα θέλαμε επίσης περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την κατανομή των πόρων ανάμεταξύ των τομέων και αναμεταξύ των προγραμμάτων και σε μια περίπτωση επίσης κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή της βοήθειας. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για το κατά πόσο οι προτινόμενες δράσεις θα συμβάλλουν πράγματι στη μείωση της φτώχεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίσαμε ορισμένα θέματα συγκεκριμένα για συγκεκριμένε χώρε. που πιστεύαμε ότι δεν είχαν ε, ε, εξεταστεί, από, αντιμετωπιστεί σωστά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν μας απάντησε. Μόνο μια φορά λάβαμε μια περιορισμένη έκτασης απάντηση για το πρόγραμμα της Κάμπια. Γι' αυτό σας ρωτώ, σας ζητώ μάλλον, ε, κύριε Επίτροπε, να φροντίσετε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ομάδας εργασίας ΣΥ. Είναι σημαντικό να έρχονται οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δίνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών ε, λαών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω και πάλι αξιότιμε κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ωστόσο είναι κάπως καταθλιπτικό όταν προσπαθεί κανείς να δει πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που είναι στο κάτω-κάτω των φορολογουμένων. Κάνουμε την προσπάθεια αυτή και τελικά έχουμε πολύ λίγες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή δεν λαμβάνονται καν υπόψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου όπως στην περίπτωση της Ερυθρέας. Όπως είπε όμως και η κυρία Ζαμπόρσκα, ε, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, και εγώ είμαι στην ομάδα εργασίας ΓΑΜΑ και έχουμε παρόμοια ε, πράγματα στη λίστα μας, ε, είναι και πάρα πολύ σύντομες οι προθεσμίες και καθιστούν αδύνατο το έργο μας. Δεν μπορούμε να εργαστούμε με χρήσιμο τρόπο. Θέλω να συμπληρώσω ακόμη κάτι. Εμπιστευτικότητα των εγγράφων. Ήδη τέθηκε αυτή από ορισμένου άλλους. Καμιά φορά μάλιστα πρόκειται για αντίφαση, διότι συντάσσουμε εκθέσεις για πράγματα και για τα οποία έχουμε συζητήσει στην Scrutiny Group για χώρες που θα έπρεπε να είναι εμπιστευτικέ οι εκθέσει αυτές αλλά οι εκθέσει που κάνουμε τελικώς είναι δημόσιο χαρακτήρα. Άρα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα της εμπιστευτικότητας των εγγράφων. Όλα τα άλλα σχόλια που ήθελα να πω έχουν ήδη καλυφθεί. Έχω ωστόσο μία ερώτηση ακόμη που ω τώρα δεν την άκουσα. Συμφωνία Κοτονού. Αυτή λύγει το 2020. Οι συζητήσει για το τι θα την αντικαταστήσει έχουν ήδη αρχίσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο 2015 εξέδωσε πράσινη βίβλο. Έγινε μετά και δημόσια διαβούλευση, η οποία έδειξε τον Δεκέμβρη. Θα ήθελα να μάθω εάν έχετε ήδη συλλέξει κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα ή κάποιες αξιολογήσεις και προς ποιαν κατεύθυνση κινούνται οι σκέψη σας για την συνέχεια και πότε σκοπεύετε να υποβάλλετε τη λευκή βίβλο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζωκίμ Σάλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, να πω λίγα λόγια από την σκοπιά της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού για τα όσα συζητήθηκαν ως τώρα. Ο κύριος Ντέβα αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο εργασίας της ε, Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, το οποίο υπάρχει ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου. Η ΔΕ Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού έχει χρέος ε, να το συντάξει το έγγραφο αυτό. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για το ότι αρχίζει αυτό με την αξιολόγηση των δράσεων της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Οι ε, επικεφαλής προσώπιών στις διάφορες χώρες μέλη λαμβάνουν την εντολή να παρακολουθούν και την χρήση και διάθεση των ε, χρημάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως, όπου γίνεται πολιτική αναπτύξεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν συμφωνίες ε, πολιτικής γειτονίας, να τα διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά μάλιστα οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών και τους ζητούμε αναέτος να υποβάλουν εκθέσεις. Αυτές οι εκθέσεις μας έρχονται από το 2012 για τον τομέα της ε, αναπτυξιακής εργασίας και από το 2015 θα μας έρχονται ελπίζω, για το 2015 και μετά δηλαδή, και για την ε, πολιτική γειτονία. Οι εκθέσεις αυτές βασίζονται σε ένα κατάλογο 16 κριτηρίων Εκεί σημειώνεται η πρόοδος διαθέσεως των ε, πόρων που διατίθεται για την αναπτυξιακή συνεργασία και από την άλλη μεριά γίνεται και μια εκτίμηση αν δηλαδή επιτυγχάνονται όντως οι προβλεπόμενοι στόχοι από τα διάφορα έργα. Αν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ή εάν οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά μεγάλοι σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Άρα από τη μια μεριά λοιπόν η δαπάνηση των χρημάτων, από την άλλη η επίτευξη των στόχων. Αυτά τα στοιχεία τα λαμβάνουμε από τις διάφορες αντιπροσωπείες της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Οι εκθέσεις αυτές λοιπόν είναι πρώτη φορά και για την απαλλαγή του προπολογισμού 2014 έκανε η Γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού ένα ε, τιτάνιο έργο να τα συγκεντρώσει τα, στοιχεία αυτά, να κάνει τη σύγκριση με τα δεδομένα του 2013 και από αυτά όντως προκύπτουν συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο εκθέσεων που θα πρέπει κάπως να μας ανησυχούν διότι αναφέρεται μέσα στα κείμενα αυτά ότι για τα RAL, για τα ρευστοποιητέα ας πούμε υπόλοιπα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό το οποίο μεταβαίνει από χρόνο σε χρόνο και δεν μπορεί απλώς να αγνοηθεί. Για 805 έργα τα οποία είναι περίπου το 50% του συνολικού ποσού της ε, αναπτυξιακής βοήθειας έχουμε κίτρινο φως, η πορτοκαλί φως αν θέλετε, όπως θέλετε, σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις πληρωμών, της τάξης του 20% του Budget Support Actions, για τα οποία πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, οι προβλεπόμενοι στόχοι, δεν είναι άλλωστε και ε, εμπιστευτική έκθεση, είναι δημόσιο κτήμα, ε, είναι ανοιχτή σε όλους. Τα συζητήσαμε αυτά με την ύπατη εκπρόσωπο στην ε, συνάντηση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολισμού. Η ύπατη εκπρόσωπος είπε όμως ότι δεν είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μαζί της, διότι αρμόδιοι για τον προϋπολογισμό δεν είναι ίδια. Είναι οι επίτροπη ΔΕΦΚΟ και ΕΚΟ, αυτή που είναι αρμόδιοι δηλαδή για ε, τα θέματα αυτά. Αυτά ρυθμίζονται και στη βάση κανονισμού. Όπως είπα, άμεσα αρμόδιοι είναι ε, οι δύο επίτροποι που προανέφερα. Αυτό είναι σημαντικό διότι και οι συνάδελφοί μας που συμμετέχουν στις διάφορες ομάδες εργασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα είπαν αυτά, ότι επιτέλους πρέπει δηλαδή η αναπτυξιακή πολιτική να ξεφύγει πια από αυτή την εντύπωση που δίνει ότι πρόκειται για ε, μια μαύρη τρύπα που ε, είναι άγνωστο τι περιέχει. Είπαμε ότι πρέπει να είναι θετικά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, τώρα όμως η πολιτική της αναπτύξεως δεν είχε βρεθεί ποτέ στο προσκήνιο της πολιτικής δράσεως. Βλέπουμε τώρα όμως πολλούς ανθρώπους από τις χώρες όπου χορηγούμε αναπτυξιακή βοήθεια να εγκαταλείπουν τη χώρα τους διότι λένε ότι δεν μπορούν για διαφόρους λόγους να θεωρήσουν ότι η ύπαρξή τους εκεί είναι ασφαλής και προσπαθούν να φάσουν στην Ευρώπη. Και όταν λέμε εμείς αναπτυχθεί η πολιτική, μιλούμε και για καταπολέμηση των ε, αιτίων αυτών που οδηγούν τον κόσμο στη μετανάστευση, στη ρίζα τους. Μιλούμε τώρα για εμπιστευτικά έγγραφα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Εγώ είδα πολλά από τα έργα ή τα προγράμματα αυτά να τα υλοποιούμε με συνεργασία με εταίρους που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. οργανώσεις των Ενωμένων Εθνών, συνεργασία με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα που χρηματοδοτούμε, συγχρηματοδοτούμε και έργα τους. Βλέπω να συνεργαζόμαστε και με άλλες χώρες ή οργανώσεις χωρών όπως η Αφρικανική Ένωση. Εφόσον χορηγούμε τα χρήματα αυτά από τα διάφορα ταμεία και μάλιστα είναι και διαφορετική η διαχείριση του ε, EDF πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και νομίζω ότι Αυτά θα πρέπει να τα συζητήσει η Επιτροπή Αναπτύξεως μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο καθένας από τη σκοπιά του. Αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε. Νομίζω μάλιστα ταυτόχρονα ότι τώρα που συζητούμε για ενδιάμεση επανεξέταση, mid-term review, πρέπει επιτέλους να εντάξουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως στον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Έχει έρθει η ώρα πια. Thank you. just to say that we are, we σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα σημείο επί του προϋπολογισμού αργότερα και θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Το είχαμε συζητήσει και με τους συντονιστές. Δηλαδή... Αλλά αυτό που συζητούμε σήμερα είναι τα θέματα του προγραμματισμού προτού δηλαδή δοθούν οι πιστώσεις. Ίσως καλό θα ήταν να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και μετά. Δηλαδή να δούμε τον αντίκτυπο και βεβαίω έχετε απόλυτο δίκαιο, έχουμε ενδιάμεση ε, αναθεώρηση δημοσιονομικών και πρέπει να δούμε πώς πάνε τα παραδοτέα, πώς πάνε τα πράγματα, τα προγράμματα και οι δράσεις που έχουμε χρηματοδοτήσει. Γιατί βλέπουμε ότι οι κονδύλια κινούνται προς διαφορετικές ε, κατευθύνσεις, έχουμε διάφορες πιέσεις και επίγουσες ανάγκες και νομίζω ότι με την ενδιάμεση αξιολόγηση θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά. Επίτροπε, είχατε πάρα πολλές ερωτήσεις. Σας δίνω μέσα το λόγο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Επιτρόπος. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τις ε, παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις. Σε διάφορα θέματα που είναι πολύ σημαντικά σχετικά με την ανάπτυξη και τις ε, πολιτικές συνεργασίας για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προκειμένου αυτές οι πολιτικές και αυτή η συνεργασία να είναι πιο αποτελεσματική. <clears throat> Εντός δηλαδή του γενικότερου πλαισίου των βιωσίμων αναπτυξιακών στόχων. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω με ας το πούμε έτσι, την αποτελεσματικότητα της γενικότερης πολιτικής ανάπτυξης Κομισιών Γιατί στα μέσα ενημέρωσης υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα όχι με την έκθεση της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου, αλλά με κάποιες διαρροές επί του από μάλλον το αναλυτικό έγγραφο της Επιτροπής το οποίο οδήγησε τα μέσα ενημέρωσης στο συμπέρασμα ότι ότι τα μισά από τα πράγματα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνουν, το δρόμο τους ή πετιόνται στον κάλαθο των αχρήστων. Δηλαδή αυτό, είπαν, αυτό είπε ο τύπος. Υπήρξε ένα εσωτερικό έγγραφο από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου που ήταν μια εσωτερική έκθεση management. Δεν ήταν μια έκθεση αξιολόγησης της συνολικότερης αποτελεσματικότητας των αεροαϊκών προγραμμάτων, αλλά με ένα ετήσιο εργαλείο διοίκησης το οποίο ε, ταυτοποιεί δυνητικές δυσκολίες και δυνητικές καθυστερήσεις ή στον κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους. Την ώρα που τα προγράμματα αυτά τρέχουν. Πρόκειται για μία απεικόνηση, στιγμία απεικόνηση του πώς έχουν τα πράγματα με τα πράγματα που τρέχουν. Και το εργαλείο αυτό, το εσωτερικό αυτό εργαλείο διοίκησης μας βοηθά να αναλαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα όταν ακριβώς επιβεβαιώνονται τα οποιαδήποτε προβλήματα. Μέτρα ώστε να επαναφέρουμε τα προγράμματα στην βέλτιστη διαδικασία υλοποίησης. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο έγγραφο να λαμβάνεται ως έκθεση για την τελική αξιολόγηση και το τελικό πόρισμα των προγραμμάτων ανάπτυξης με τις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και την τυχόν συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς, ε, με τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς. Έχουμε τη Δημοσιονομική Επιτροπή, έχουμε τους ελεγκτές, τακτικές εκθέσεις από όλους αυτούς τους συναρμοδίους και η, πρέπει να σας πω ότι ε, τα ποσοστά λάθους βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα από προγράμματα που εμφαρμόζονται εντός του εσωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσωτερικά, in-house που λέμε. Παρά το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε για τα προγράμματα ανάπτυξης. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι καινούριο, για κάτι εξαιρετικό, για κάτι ευνηδιαστικό. Κάθε χρόνο έχουμε ενδείξεις για τα προγράμματα εκείνα που μπορεί να καθυστερήσουν, που μπορεί, μπορεί λέω, να συναντήσουν την οποιαδήποτε δυσκολία και αυτό ε, περιγράφεται σε αυτό το εσωτερικό εργαλείο. Δεν μπορεί αυτό να θεωρείται αξιολόγηση συνολική των προγραμμάτων. Το καλύτερο εργαλείο θα ήταν εδώ στην Επιτροπή των Δημοσιονομικών Θεμάτων και στο ελεκτικό συνέδριο θα ήταν τα κατάλληλα βήματα ώστε να αξιολογείται η τελική εν πάση περιπτώσει επίδοση των προγραμμάτων μας. Και θα ήθελα να εστιαστούμε σε, στα πραγματικά γεγονότα από το πλαίσιο αποτελεσμάτων. Results framework, λέει ο Επίτροπος. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να θεωρείται βάση ε, προκειμένου να αξιολογούνται τα παραδοτέα, τα αποτελέσματα τελικής επίδοσης των προγραμμάτων και όχι σε κάποια ενδιάμεση φάση. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, θα έλεγα ότι το έγγραφο που κυκλοφόρησε και που εξετάστηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής και όταν εξηγήσαμε μπάστε τόσοι όλες τις σχετικές λεπτομέρειες βασίζεται το δημοσίευμα δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης βασίζεται σε μια τελείως λανθασμένη υπόθεση εργασίας ότι εφόσον υπάρχει μια οποιαδήποτε ένδειξη κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος αυτό είναι καταδικασμένο να αποτύχει, δεν είναι καθόλου έτσι. Έχουμε ένα κύκλο ζωής των προγραμμάτων στα έργα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και μερικέ φορέ χρειάζεται και πάρα πολλά χρόνια, 27-30 χρόνια. Δηλαδή αυτά μάλλον που γράφτηκαν για τα 27 με 30 χρόνια δεν βασίζονται επί τη βάση πραγματικών έργων ή προγραμμάτων. Εμείς είχαμε 5 με 6 χρόνια κατά μέγιστον ως απαραίτητο χρόνο που θα χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Δεν είναι μέσο όρο αυτό που σα λέω, αλλά είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλα τα μέλη της Επιτροπής εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Κομισιόν στις ε, αρμόδιες υπηρεσίες να εργαζόμεθα επί των στοιχείων που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο αποτελεσμάτων που θα είναι το μόνο εργαλείο που θα μπορέσει να μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την τελική επίδοση των προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Επίτροπος. Να επανέλθω τώρα στην υλοποίηση του στρατηγικού διαλόγου υπό το DCI και την παρακολούθηση του EDF. Να ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας ε, τις επικοδομητικές σχετικά με την ε, όλη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα δούμε ως στοιχεία από τα οποία πρέπει να δουλέψουμε από κοινού για να προοδεύσουμε. Ε, σε γενικέ γραμμέ η συνεργασία της Ετροπή ΔΕΒΕ και της Κομισιόν οι ε, κοινέ προσπάθειες αυτές είναι και υπήρξαν υψηλωτά του επίπεδου σε αυτό τον πρώτο χρόνο ε, εντολής και για την Κομισιόν και για την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Υπάρχουν θέματα ή στα πλαίσια της διαθεσμικής συνεργασίας των σχέσεων των θεσμικών αλλά δεν θα έπρεπε κανείς να το βλέπει ως ε, μια αντιπαράθεση εξουσίας για το ποιο θα πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος μας και η συνεργασία μας πάντα κατευθύνεται από τον ενθουσιασμό, την φιλοδοξία, την εμπειρογνωμοσύνη και την βούληση κοινή συνεργασίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο προκειμένου να επιτύχουμε, να εκριζώσουμε την ένδια και να εκπληρώσουμε γενικώ τους στόχους της ιεραϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας. Uh, οι οποίοι στόχοι βεβαίως κατευθύνονται και πλαισιώνονται από την διαθεσμική συμφωνία συνεργασίας, αλλά ιδιαίτερα στην, στο πεδίο αυτό, στην περιοχή αυτή, υπάρχει το περιθώριο να κυριθούμε εντός του πλαισίου, εντός των ορίων αυτών, αποτελεσματικότερα. Προκειμένου να έχουμε περισσότερες πληροφορίες διαθεσή μας περισσότερη γνώση ώστε να ε, βοηθήσουμε στην καλύτερη συνολική επίδοση της συνεργασίας μας. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω αμφότερες τις υπηρεσίες μας να κινούνται εντός του πλαισίου βεβαίως της διαθεσμικής μας συνεργασίας και διευθετήσεων και με το κοινό συμφέρον που έχουμε ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών και στον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα μας επέτρεπε και εγκαίρως να αποστέλουμε τα έγγραφα Uh, uh, uh, and να έχουμε δηλαδή την καλύτερη να τηρούμε, την καλύτερη δυνατή διαδικασία παρακολούθησης ε, και να εξασφαλίζουμε και την ε, έγκαιρη και τακτική προσέλευση των εκπροσώπων της Κομισιόν στα, στις συναντήσεις της ομάδος, των ομάδων εργασίας. Ε, γιατί μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε νομίζω να υπερκαλύψει και να διορθώσει τα όποια στοιχεία και ελλείψεις εσείς επισημάνατε. Εμείς νομίζω ότι έχουμε καταδείξει την ε, διαθεσιμότητά μας να πάμε μέχρι τα όρια, τα όρια λέω, των διαθεσμικών αυτών διευθετήσεων συνεργασίας. και σε σχέση με την άτυπη παρακολούθηση του EDF την οποία απεδέχθημεν και επαναλάβαμε την δέσμευση και του... Εγώ ο ίδιος επαναλάβα τη δέσμευση του προκατόχου μου. Εκφράζοντας τη βούλησή μου να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επί των προγραμμάτων αυτών ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν οι σημερινές αυτές τις συζητήσεις να είναι πραγματικά εφαλτήριο για τις ε, υπηρεσίες μας σε αγαστό πνεύμα συνεργασίας ώστε να καλύψουμε αυτά τα στοιχεία που επισημάνατε σήμερα για τις διαδικασίες ε, παρακολούθησης ε, και για το πώς μπορούμε καλύτερα να συνεχίσουμε, ξαναλέει ο Επίτροπος. Επίσης να αναφερθώ στο θέμα της συνολικής δυνατότητος υλοποίησης και συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύτερο, στο παγκόσμιο πλαίσιο της, ε, του θεματολογίου 2030. Έχουμε θέσει την προσέγγιση της συνολικής ομπρέλας σχετικά με αυτές τις έννοιες ε, της ευρύτατης ερμηνείας και εφαρμογής ε, παγκόσμιος κλίμακας και εντός και εκτός και στις εξωτερικές μας δράσεις σχετικά δηλαδή με τους στόχους αυτού του θεματολογίου 2030 και πολύ σύντομα θα Είμαστε έτοιμοι με ένα ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο που δεν θα είναι απλώς η στρατηγική ανάπτυξη και απασχόληση για την Ευρώπη 2030, αλλά θα ενσωματώνει την έννοια της βιωσιμότητας σε όλες αυτές τις πολιτικές προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να έχουμε αυτή τη στρατηγική προσέγγιση προς την εφαρμογή της, ε, του θεματολογίου 2030. Ανεξαρτήτως της ταχύτητος βεβαίως αυτού του Sustainable Europe 2030, ας το ονομάσουμε έτσι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως θεματολογίου, θα πρέπει από κοινού να συνεργαζόμαστε ώστε να ορίζουμε καλύτερα τις εξωτερικές μας δράσεις, τις συνεισφορές μας ή τις πολιτικές ανάπτυξης για τις χώρες εταίρους. Και πρέπει λοιπόν να επανεξετάζουμε και να αναθεωρούμε την ευρωπαϊκή συνένεση επί των θεμάτων ανάπτυξης που θα πρέπει να έχουμε προκειμένου να έχουμε μια πολιτική και προσέγγιση όσο πιο συνεπή γίνεται. Και αντί να έχουμε 29 διαφορετικές πολιτικές ε, υλοποίησεις για το κάθε κράτος μέλος και για την ε, Κομισιόν, να έχουμε μία συνέντευξη, λοιπόν για τα θέματα ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Και πρόκειται για μια περιοχή στην οποία είχαμε μια αρχική στήριξη στα κράτη-μέλη τον περασμένο Δεκέμβριο στο άτυπο ε, Συμβούλιο Ανάπτυξης ότι θα πρέπει να εργαστούμε σε μια αναθεωρημένη συνένεση για τα θέματα ανάπτυξης και νομίζω ότι φέτος θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο για να έχουμε αυτήν την αναθεωρημένη συνένεση μέχρι το τέλος του έτους. Uh, also, uh, Και αυτό βεβαίως σχετίζεται και με την, ε, με την όλο σχεδιασμό μετά την Κοτονού ή εν πάση να την πούμε την post-2020 περίοδο με τους εταίρους ΑΚΕ είχαμε ξεκινήσει μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης, τώρα ολοκληρώθηκε αυτή και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πρώτη άποψη, συνολική άποψη, έποψη όπως λένε κάποιοι, αυτής της όλης διαδικασίας. Και μέχρι το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε και τον, την ανάλυση αντικτύπου για τα διάφορα δυνατά σενάρια της ευρωπαϊκής ε, ανταπόκρισης προς την περίοδο μετά την Κοτονού. Και νομίζω ότι αυτήν την εποχή του χρόνου θα έχουμε σαφείς θέσεις και προτάσεις προκειμένου αυτές να συζητηθούν με τους εταίρους μας σαφώς πριν από το 2018 που θα είναι και το εναρκτήριο έτος των συναντήσεων post κοτονού οι οποίες συναντήσεις θα πρέπει να τεθούν και στο πλαίσιο της ε, συνεισφοράς προς την, ε, το θεματολόγιο 2030 και προς το, <clears throat> την αναθεωρημένη συνένεση για θέματα ανάπτυξης που ανέφερα νωρίτερα. Τα σχόλιά σας σχετικά με τις ε, επιχειρήσεις Trust Fund δεν θα αποκαλούσα αυτές τις, αυτά τα εργαλεία ή αυτή την προσέγγιση τόσο καινοτόμα Ναι, έχουμε τρία διαπιστεύματα δημιουργήσει Αφρικής, Μαντά για χώρες Συρίας και τα θέματα μεταναστών κτλ. Και, και το τρίτο το πιο φιλόδοξο το Ευρωπαϊκό Trust Fund για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ε, της μετανάστευσης στην περιοχή Σαχέλ και του και εξετάζουμε και τη δημιουργία ενός ακόμα για την Κολομβία εφόσον ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Η βασική, ο βασικός λόγος της ύπαρξης των, καταπιστευμάτων αυτών είναι ότι ο κύκλος ζωής των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων είναι όπως σας είπα νωρίτερα 5 με 6 χρόνια ενώ εδώ μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την άμεσα, να έχει τον άμεσο αντίκτυπο εντός ενός δύο ετών το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση των ε, επιπτώσεων ε, των μεταναστευτικών ροών, ε, για τα θέματα απασχόλησης ε, και στις χώρες προέλευσης και στις χώρες διαμετακόμισης των μεταναστών και της ευελτίωσης της δυνατότητός τους να αντιμετωπίζουν, να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματα μεταναστευτικών ροών. Θα συνεχίσουμε με τα καταπιστεύματα, αλλά δεν θα θέλαμε να είναι απλώς ένα νέο ε, front loading των υφισταμένων αφρικανικών μέσων που είχαμε γιατί είχαμε προκειμένου να επιτύχουμε το 1,8 δις ε, που είχαμε για τα συνολικά ως πόρους ανάπτυξης είχαμε διάφορα μέσα αναπτυξιακά και περιμένουμε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν το αντίστοιχο ποσό, προς το παρόν απέχουμε πολύ. Μόνο 83 εκατομμύρια, αν ακούσαμε καλά. Είχαμε από τα κράτη-μέλη και κάποιους άλλους δωρητές. Προκειμένου λοιπόν αυτά ε, τα καταπιστεύματα να είναι συνολικότερης εμβέλειας και πιο διεθνούς ενδεχομένως εμβέλειας Κάπως έτσι βλέπουμε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε ε, Δεν φαντάζομαι όμως ότι αυτό το μέσον θα καταστεί ε, ο μόνος ή ο βασικότερος τρόπος παρέμβασής μας, το καταπίστευμα. Δεν φαντάζομαι Ακόμα και το μεταναστευτικό καταπίστευμα για την Αφρική, όπως σας είπα το 1,8, είναι πολύ μικρότερο από τη συνολική δέσμη παρέμβαση στην Αφρική, τη δική μας που είναι 20 δις. Απλώς θα είναι συμπληρωματικές δράσεις που θα τρέχουν παράλληλα με, την ε, τακτική χρηματοδότηση, με τα τακτικά κονδύλια. Και θα ήθελα να σας βεβαιώσω πραγματικά ότι ετούτη η Κομισιόν και εγώ ιδιαίτερα ως επικεφαλής θεμάτων διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας το σύνολο του εύρους του πλαισίου της διαθεσμικής μας συνεργασίας για τα θέματα αυτά και είμαι βέβαιος και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και θα τα καταφέρουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές διευθετήσεις ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις δικές σας παρατηρήσεις εις τον ύψιστο δυνατό βαθμό και καλύτερα και από πριν ή δυνατόν. Για τις διαδικασίες λοιπόν άτυπου διαλόγου και παρακολούθησης θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να έρχομαι σε τακτική βάση, σε όποια βάση, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε αυτό καλύτερα να συνεισφέρει σε στο καλύτερο δυνατό κοινό impact, αντίκτυπο επί των προγραμμάτων. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αν θέλετε κάτι πολύ σύντομα, πρώτα εσείς. Όχι άλλες ερωτήσεις. Εκτιμώ πολύ τους δύο συναδέλφους μας, τον ε, αντιπρόεδρο μας κύριο Ντέβαλα και τον κύριο Τσέλερ Όμως εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, Αναπτύξεως ήταν στη συνάντηση με την κυρία Μογκερίνη, αλλά δεν μας έδωσαν το λόγο. Τώρα, για αυτό το λεγόμενο έγγραφο εργασίας το οποίο δημοσίευσαν ε, και οι Sunday Times, προσοχή, βασίζονται στις αιτήσει εκθέσεις των γραφείων των ε, αντιπροσωπιών από μη κοινοτικέ χώρες και δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο μια ενσταντανή φωτογραφία, μια στιγμή φωτογραφία, όχι το τέλος ενός έργου. Δεύτερο, το έγγραφο εργασία, ή μάλλον οι Sunday Times αναφέρονται σε δύο συγκεκριμένα έργα τα οποία λένε ότι είναι αμφιλεγόμενα και αποτυχημένα. Ένα στα νησιά Κομόρε για ηλιακή ενέργεια και ένα για την καταπολέμηση τη διαφθορά στην Ιγυρία. Αντίθετα όμω από ό,τι λέει το ε, έντυπο αυτή, η εφημερίδα αυτή και το έγγραφο αυτοεργασία, αυτά τα ε, προγράμματα λειτουργούν. Δεν, εγώ, εγώ δεν επιθυμώ να υπεραμεινθώ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βεβαίω υπάρχουν πολλέ παραλήψει. Αλλά όχι όμω να λέμε τέτοια πράγματα και ιδίω με τόσου πολλού παρόντε σε αυτή την ε, ε, συνεδρίαση. Εκτιμώ ιδιαίτερω του συναδέλφου μου που προανέφερα και είναι πραγματικά εξαίρετα μέλη τη Επιτροπή Αναπτύξεω, αλλά του παρακαλώ να διαβάσουν την αντίδραση της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσίευμα των Sunday Times. Πολύ σημαντική η αντίδραση αυτή, διότι αλλιώς θα πρέπει να θεωρήσουμε όλες και όλοι ότι διέρευσε το έγγραφο αυτό προς το Sunday Times για να ενισχύσει το προστάσιο αυτών που είναι υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Brexit. Charles Goerens, πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ ε, σοβαρή συζήτηση αυτή και γι' αυτό ζητώ το λόγο. Δεν θα ήθελα με συνενοχή δική μας να δώσουμε μια ασαφή ιδέα στον τύπο ότι δήθεν δεν είναι πλέον αξιόπιστη η πολιτική αναπτύξεως της Ένωσης. Δεν βλέπω απολύτως κανένα στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ μιας κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς. Τα όσα είπα εγώ είχαν την έννοια ότι αν καθυστερεί κάποιο έργο χρειάζεται να ληφθούν μέτρα προφύλαξης. Και να ε, επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου. Χωρίς όμως να υπάρξουν αυλεψίες σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του έργου. Αν κάποιο έργο χρειάζεται περισσότερο χρόνο, σημαίνει αυτό ότι πρέπει να εγγύψουμε στο πρόβλημα. Με κανένα τρόπο δεν θέλω να ε, φύγει κανείς από την αίθουσα αυτή θεωρώντας ότι εδώ επικρίνουμε την ε, πολιτική ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Πολλοί ανά τον κόσμο επιτίθενται στην αναπτυξιακή συνεργασία. Όχι όμως να την καταρρύψουν με λόγους που δεν είναι αιτιολογημένοι. Αυτά τα λέω όχι μόνο για να μείνουμε μεταξύ μας, αλλά και για να ακουστούν και προς τα έξω. Χρειάζεται ανακοινωθέν τύπου, το οποίο να είναι σαφέστατο και αυστηρότατο είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από την Επιτροπή Εξωτερικών Δράσεων για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. μη γινόμαστε συνένοχοι μιας πραγματικής επίθεσης έξωθεν κατά της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Διότι αυτοί που τα λένε αυτά δεν ε, με εξετάζουν το θέμα όπως εμείς έχαμε τον κύριο Πίνκστιν του ελεγκτικού συνεδρίου πριν από λίγες μόνες, ε, πριν από λίγους μήνες, που μέμφεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν εκτελεί καλά τα έργα. Από την άλλη μεριά, το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο εξακολουθεί να επικρίνει τον υψηλό βαθμό συνοδευτικών δαπανών των έργων. Αλλά εδώ είτε το τελεσχεί είτε το άλλο. Και ο ΩΣΑ λέει καθαρά ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό για να εκτελεί τα διάφορα έργα ή προγράμματα. Χρειάζεται λοιπόν να εγγύψουμε στο φάκελο αυτό ώστε η υπόθεση αυτή να μην λάβει τις διαστάσεις που κανείς από εμά δεν θα ήθελε. Και το υπενθυμίζω σε όλους τους συναδέλφους μου, είτε είναι μέλη της Επιτροπής Αναπτύξεως είτε της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολισμού ότι η, Επιτροπή, η, ε, η αναπτυξιακή συνεργασία είναι από τα πλέον σημαντικά τμήματα του κεκτημένου. Μην την ρίξετε στα σκυλιά. Ευχαριστώ, Λίντα Μακάβαν σημαντικά και σοβαρά πράγματα αυτά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρό τρόπο. Ελπίζω ότι αυτά θα τα συζητήσουμε και στους συντονιστές. Μου ζήτησαν να σχολιάσω ένα έγγραφο και μετά εγώ δεν το βρήκα. Πουθενά. Διότι δεν ήταν επίσημο έγγραφο. Δεν είναι τρόπος αυτός να γίνεται η δουλειά. Να μην το συζητήσουμε άλλο κύριε Ζέλερ. Πολύ σύντομα τότε, Ιωακήμ. Μα εδώ εμφανίζει το πράγμα σαν να το βάλαμε εμείς το έγγραφο αυτό επιτάπητος. Όχι, πρόκειται για σύνοψη των εκθέσεων των αντιπροσωπιών της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Τα στοιχεία που λέει είναι σοβαρά και πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να γίνουν αλλαγές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Και ε, επίσης η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων αυτό λέει. Άλλο που συζητούμε εδώ ότι συχνά δηλαδή δεν γνωρίζουμε καν τι γίνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια. Μας στέλνουν τα διάφορα project και εχουμε τρει τρει-τέσσερι μέρε για να μελετήσουμε annual action plans, multi-annual action plans κτλ. Μετά το τι γίνεται με αυτά τα σχέδια, έχετε εσεί καμιά ιδέα. Το 2014 ζητήσαμε μια επισκόπηση για να δούμε ποια ε, έργα εγκρίθηκαν από ε, ε, ζητήσαμε ένα πίνακα Excel και μας επέτρεψε να τον δούμε μόνο σε εμπιστευτική συνεδρίαση. Μα γιατί εμπιστευτικό το έγγραφο αυτό. Χρειάζεται να είναι διαφανές, δεν χρειάζεται να είναι εμπιστευτικό, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ορθή. Σαλ Γκέρενς, απευθύνομαι στον κύριο Τσέλερ. Εγώ δεν θέλω να επιτρέψω να προκληθεί η εντύπωση ότι εδώ έχουμε απέναντί μας κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος δικαίως ζητείτε την διαφάνεια. Δεν επιτρέπεται όμως, επαναλαμβάνω, να αφήσουμε να ηγεθεί η υπόνοια κακοδιαχείρισης. Διότι αυτή αξίζει την υποστήριξη και την υπεράσπισή μας, έθεσε ό,τι αποδειχθεί το ενάντιον, εάν ποτέ. πόρο απέχουμε από την εντύπωση ότι ίσως κάτι συμβαίνει που δεν είναι ορθό. Θα συζητήσουμε βεβαίω για την απαλλαγή. Αν έχετε τροπολογίε για συγκεκριμένα θέματα που θα πρέπει να λάβει υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο, τότε εξετάστε τα έγγραφα, κάντε τι τροπολογίε και θα τι συζητήσουμε με την ευκαιρία αυτή. Και για τα θέματα τη ε, διαφάνεια και του έχω, θα τα κάνουμε αυτά το ίδιο στον προγραμματισμό μα. Σήμερα θα δούμε πώ θα βελτιώσουμε την επεξεργασία των ε, θεμάτων. Έχετε τρόπο να κάνετε τις προτάσεις σας, συζητήστε με τις πολιτικές ομάδες και κάντε το σχεδιασμό σας. Ευχαριστώ επίσης και τον Επίτροπο που έμεινε μάλιστα κοντά μας πολύ περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί και περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας. Ας είναι μάλλον το 9 καλύτερα αυτό, διότι έχουμε όπως σας εξήγησα πριν τον κύριο Brian Hayes ο οποίος ε, ζήτησε να προταχθεί το θέμα του και τώρα προχωρούμε και με κάποια καθυστέρηση. Το υπαριθμό είναι 9 λοιπόν κύριοι συνάδελφοι και μετά θα πάμε στα επόμενα 6, 7, 8. Πρόκειται για συζήτηση, για μια γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πιο περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον. Και θα εξετάσουμε τις ε, πολιτικές της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Έχετε το λόγο Brian. Όσοι αποχωρείτε παρακαλώ πράξετε το ησύχω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Επαναλαμβάνω όσοι αποχωρούν από την αίθουσα να το κάνουν ήσυχα. Μην ξεκινάτε τη συζήτηση μέσα στην αίθουσα έξω. Για να ακούμε και τον ομιλητή. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ επίσης για την ε, ευελιξία σα, τη δυνατότητα που μου δώσατε να ε, παρουσιάσω την ολοδότησή μου τώρα γιατί θα πρέπει να παρευρεθώ σε ψηφοφορία στην οίκον σε λίγα λεπτά. Η γνωμοδότηση αυτή πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, ε, είναι μάλλον επί ενό πολύ σημαντικού εγγράφου Τη έκθεση που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί στι αλλαγέ που συντελούνται παγκοσμίω όσον αφορά την. Ε, ότι είμαστε ο κόσμος όλο και πιο συνδεδεμένος. Αυτό που λέγεται είναι ότι πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει να δοκιμάσουμε τι θα συμβεί και σε πολλές περιπτώσεις αποτύχαμε. Ανταυτού θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας θεσμικό μηχανισμό όπου να αξιολογεί την, ε, τα μαθήματα που μπορούμε να, να, να εξαγάγουμε από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, έτσι ώστε στο μέλλον να βελτιώνουμε τις παρεμβάσει μας. Δεύτερον, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο όραμα, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε τα όλο και πιο περίπλοκα διεθνή θέματα. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται πάντα δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβει κανείς ποιες είναι οι επιδιώξεις της Ένωσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουμε εσωστρέφεια, δεδομένη της μεταναστευτικής κρίσης, δεδομένης της κατάστασης σε πολλές χώρες του κόσμου, θα πρέπει να έχουμε μια ε, ε, πολιτική ως Ευρωπαίοι για να ε, συνεισφέρουμε με τα μεγάλα ποσά που συνεισφέρουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια ανά τον κόσμο. Και για να γίνει αυτό αποτελεσματικά χρειάζεται μια διαδικασία αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε στους διεθνείς οργανισμούς. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα θέματα που αναδεικνύω και στο γνωμοδέτησή μου. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της συνοχής το δεύτερο είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης των αιτιών, των γενεσιουργών αιτιών, των προβλημάτων στη ρίζα τους, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετανάστευση και τη σχέση μας με χώρες της Αφρικής. Όσον αφορά το πρώτο σημείο τώρα, τη συνεκτικότητα, τη συνοχή, πρέπει να ενισχυθεί κατά την άποψή μου. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών μας πολιτικών. Επίσης μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αυτό το αναδεικνύω στην εκθεσή μου ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να ε, καταφέρουμε να έχουμε τη συνοχή που επιθυμούμε, να είναι ξεκάθαρο και στα 28 κράτη-μέλη τι επιθυμούμε και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων είναι συγκεκριμένος και κρίσιμος. Επίσης, η επιδίωξη των αναπτυξιακών στόχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της όσον αφορά τώρα τους, στόχου τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να, να, να τηρούνται, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, καλή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά προβλημάτων που μας απασχολούν έντονα όπως η μετανάστευση. Θα πρέπει να να αντιδρούμε στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται γρήγορα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να προσαρμόσουμε το πλαίσιο με το οποίο παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει αυτό πιο ταχύ. Επίσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την σημασία και τις δυνατότητες που μας, δίνουν, μας δίνονται εάν και τα 28 κράτη-μέλη λάβουμε από κοινού δράσεις. όχι μόνο για τη βελτίωση της κατάστασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και για την βελτίωση της κατάστασης σε άλλες περιοχές του κόσμου. Τονίζω λοιπόν τη σημασία της υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων, καθώ επίση και τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου κτλ. Και το τρίτο σημείο που ε, ήθελα να δείξω, τη σχέση μας με την Αφρική, θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική μας όσον αφορά τη μετανάστευση, το εμπόριο και την ασφάλεια. Το 2020 λίγη η ε, η συμφωνία για τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ και θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα τη συνεχίσουμε δεδομένων των κοινών μας ε, στόχων, επιδιώξεων και συμφερόντων. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που θα ήθελα να δείξω σχέση με τη στρατηγική μας για τα, για επόμενα χρόνια. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών τροπολογιών είναι μέχρι την Παρασκευή και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που θα μου υποβληθούν με τη μορφή τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κάποιος συναδελφός το λόγο. Ο κύριος Φροντζούλητ. Είμαι σχεδόν συζητητής για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση είναι καλή, έχει συνταχθεί καλά και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι τονίζεται το θέμα της συνοχή. Και ότι λέγεται ότι θα πρέπει να, να ε, βελτιωθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των, εσω, των πολιτικών στο εσωτερικό της Ένωση και τη εξωτερική δράση. Επίσης, πιστεύω θα έπρεπε να βελτιωθεί και ο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων και με τα κράτη-μέλη και με τα κοινοβούλια. Προστηρίζω επίσης την ιδέα ότι η αναπτυξιακή βοήθεια, οι πολιτικές για την ανάπτυξη είναι το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ρίζα του σε όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, κόσμο των προβλημάτων ασφάλειας, των προβλημάτων μετανάστευσης. Αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες. Διαφορετικά ε, θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο ζωή μας εάν συνεχίσουν να κλιμακώνονται οι συγκρούσεις και αν αυτό οδηγεί σε όλο μεγαλύτερε μεταναστευτικέ ροέ προ την Ευρώπη. Αναφέρεται επίση και το υποστηρίζω μια ευέλικτη χρηματοδότηση η οποία να αντιμετωπίζει και τα ζητήματα ασφάλεια όταν αυτά συνδέονται με την ανάπτυξη. Υποστηρίζω επίσης την προσπάθεια να προσαρμοστούμε, να προσαρμόσουμε τον τρόπο υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων στη νέα πραγματικότητα. Ε, πολλά θετικά στοιχεία έχει αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η έκθεση, θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα. Θα περιοριστώ σε αυτά. Απλώ θα ήθελα να συζητήσω, κυρία Πρόεδρε, γιατί και εγώ πρέπει να φύγω για άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια και ήμουν εισηγητής ε, και για το θέμα ε, των ε, Σαλίας και για το θέμα της απαλλαγής του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να συζητήσω να μου δώσετε το λόγο να τα παρουσιάσω αυτά τα θέματα και να φύγω γιατί θα πρέπει να φύγω. Η κυρία Μακάβαν. Ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τελειώσουμε ώστε να το πιο γρήγορα. Έχω έναν, άλλο ακόμα έναν ομιλητή και μετά θα συζητήσουμε το θέμα της απαλλαγής. Μαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό <clears throat> που πρώτο θέμα έρχεται στην έκθεση η συνοχή πολιτικής. Εκεί χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμη. Και στην εσωτερική, δηλαδή συνοχή, αλλά και στην συνοχή προ τα έξω, στην διάσταση προ τα έξω. Για παράδειγμα, για αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχεια. Οι συμφωνίε μα για την αλία, οι περιορισμένες προσπάθειες στην αντιμετώπιση των ε, ε, παράνομων διακινήσεων χρήματος έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις χώρες που βρίσκονται στον δρόμο της ανάπτυξης και έχουν τελικά ως αποτέλεσμα μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς εμάς. Δεν είναι δυνατόν χρήματα που δίνονται για την ανάπτυξη να δαπανώνται για άλλους σκοπούς εκτός από την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης. Είχαμε δώσει χρήματα το 2014, 2,9 εκατομμύρια για παράδειγμα μέσω του DCI για την προστασία των συνόρων της Λιβικής Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν τα χρήματα αυτά να μην δίνονται για την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά για λόγους ασφάλειας, για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας. Οι στόχοι των Ενωμένων Εθνών <clears throat> για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη για μέχρι το 2030 επίσης πρέπει να αναφερθούν στην έκθεση. Ζητήματα ασφάλειας και ειρήνης αποτελούν απόσπαστο μέρος της προσπάθειας αυτής. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, είναι σημαντικό να τονίσουμε και ότι και τα Ηνωμένα Εθνή και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να οργανωθούν με πιο δίκαιο τρόπο, ότι πρέπει να είναι δικαιότερη και αντιπροσώπευση των φτωχότερων χωρών. Και βεβαίω πρέπει να είναι δικαιότερη και η στόχη πολέμηση τη φτώχεια. Αυτά. Σα ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Μήπω θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Σύντομα, μια και θέλει να φύγει και ο εισηγητή και ο ηγητή. Μπράιαν, έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, απλά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους θα ήθελα. Που πήραν το λόγο. Περιμένω τις τροπολογίες τους. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να μην ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για ένα πλαίσιο, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των πολιτικών μα ήδη από το πλαίσιο, το γενικό πλαίσιο. Και μετά να δούμε πώ αυτό εξειδικεύεται στην πράξη. Πράγματι, τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα φάνηκε ότι αυτό ακόμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η απαιτούμενη συνοχή στι πολιτικέ μα. Την οποία παρόλα αυτά έχουμε συμφωνήσει. Ε, Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ αυτέ οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, τοποθετούνται στη διεθνή κοινότητα πώς δραστηριοποιούνται για παράδειγμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και πώς εμείς θα τις υποστηρίξουμε σε αυτό. Είναι σίγουρο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί του πλαισίου, το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ε, ευρύ, ε, γενικό, μια και μιλούμε για το σύνολο των πολιτικών της Ένωσης και το σύνολο των στόχων μας. Η πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 29 Ιανουαρίου, δηλαδή την Παρασκευή αυτή. Βεβαίως σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή για την Ανάπτυξη ΔΕΒΕ να περιοριστεί στις αρμοδιότητες της δεδομένου ότι επί της ε, ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η αφέτη εξωτερικών υποθέσεων. Αυτό θα βοηθήσει και τον ε, εισηγητή έτσι ώστε τελικά να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση η οποία θα έχει αντίκτυπο, θα επηρεάσει τα πράγματα. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στις δύο επόμενες, ε, δύο επόμενα θέματα. Έχουμε δύο ξεχωριστές εκθέσεις στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για το DCI αφενός και για το EDF. Ε, ο εισηγητής είναι ο κ. Σοντζόλητσα, μιας και μας είπατε ότι πρέπει να φύγετε, έχετε αμέσως τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σε το EDF, το Ταμείο Καλωσορίζω την δημιουργία των ειδικών ταμείων για τη Συρία και για την Αφρική, αλλά επίσης κρώ τον κόδωνα του κινδύνου για το γεγονό ότι ε, χρησιμοποιούνται ποσά από την ανάπτυξη, που ήταν για την πολιτική ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση των, των προσφυγικής κρίσης. για να φροντίσουμε χρήματα για την αναπτυξιακή συνεργασία να μην πηγαίνουν σε τομεί πολιτική που δεν αφορούν πραγματικά την αναπτυξιακή συνεργασία, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση, μια, μια ε, μελέτη. Έχουμε δεσμευτεί ότι το 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο θα πηγαίνει σε άμεση αναπτυξιακή συνεργασία και στο επίπεδο τη Ένωση και στο επίπεδο των κρατών μελών. Αυτό το χαιρετίζουμε. Βέβαια, θα πρέπει η χρηματοδότηση ε, των ταμείων για την κλιματική αλλαγή και άλλων ταμείων να είναι επαρκής, παρά την σημασία που έχουν οι γενικές πολιτικές, είναι εύκολο κανείς να ποσοτικοποιήσει και να, να ελέγξει ποια ήταν τα, ποσοτικά αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχάμε και τη σημασία ποιοτικών δικτών, όπως για παράδειγμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο, σε ειδική του έκθεση, έχει αναφέρει ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγονται τα χρηματοδοτούμενα project θα πρέπει να γίνουν πιο σαφή και το υποστηρίζουμε αυτό επίση. Ο κύριο Στία και μετά η κυρία Χόιμπρουκ. Κύριο Στία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, <clears throat> καθότι ο συνάδελφο πρέπει να φύγει, ήθελα να θίξω το θέμα του σχετισμού μεταξύ της ανάπτυξης και των θεμάτων ασφαλείας. Αυτό το αναφέρετε κι εσείς και αποτυπώνετε στα έγγραφα. Έχοντας λοιπόν εγκρίνει ε, μια νέα δέσμη στόχων, έχουμε g 16 σχετικά με τις δικασίες ειρήνευσης και αν δεν ε, απατώμε υπάρχει από τον ΩΣΑ ένας νέος ορισμός ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και την χρηματοδότηση που θα σχετίζεται με τα θέματα ασφαλείας. Και φαντάζομαι ότι θα είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων από αυτού και τουλάχιστον από τη δική μας μεριά αυτό το υποστηρίζουμε. Η πρόθεσή μας λοιπόν θα είναι να αποτυπώσουμε την ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία προκειμένου και να εφαρμόσουμε την FTG16 χωρίς να υποσκάπτουμε τα θέματα που τίθενται. Βεβαίως δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ε, ειρήνη. Ευχαριστώ. Και στις δύο γνωμοδοτήσεις υπάρχει ανάγκη βελτιώσεως αν πάρουμε την απαλλαγή του συνολικού προπολογισμού του 2015, το ελεγκτικό συνέδριο εκτιμά το σφάλμα σε 3,8 περίπου το 100 για το ε, ε, Ταμείο Αναπτύξεως, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως, ενώ το 2014 3,4%. Άρα δεν μπορεί να δώσει θετική αξιολόγηση. Τα περισσότερα σφάλματα κατά το ελεγκτικό συνέδριο προκύπτουν από την μη τήρηση των διατάξεων για τη δαπάνηση των χρημάτων. Και κάποιοι έλεγχοι εκ των προτέρων μείωσαν το ποσοστό των σφαλμάτων. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη και καλύτερη έλεγχη πριν δαπανηθούν τα χρήματα. Παρόμοια σχόλια για το υπαριθμόν 8. Η κυρία Χάουταλα είναι αυτή που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Αλλά επειδή ο εισηγητής αναγκάστηκε να αποχωρήσει, θα καταθέσουμε τροπολογίες. και αυτές θα τις συζητήσουμε με τους κοιόδης Ναι, Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν κάτι θα ήθελα να πει. Όχι. Ήμασταν όλοι πολύ σύντομοι σήμερα. Γνωρίζουμε λοιπόν τις προθεσμίες για τις τροπολογίες που είναι Τετάρτη Τετάρτη 27 του μηνός στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Και θα επανέλθουμε τώρα στο σημείο 6 που είναι συμφωνία αλληλείας με την Γρυλανδία Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κούλογλου της Γκουε, δεν είναι εδώ σήμερα αλλά έχουμε αντικαταστάτη την Λόλα, παρακαλώ Ευχαριστώ Λίντα. Ο κύριος Κούλογλου παράγματι δεν μπορούσε να είναι εδώ και επομένως σας διαβιβάζω τη συγνώμη του και έχω αναλάβει να παρουσιάσω εγώ τη συμφωνία αυτή. Μιλούμε για μία από τις 27 χώρες της περιοχής 4 της συνθήκης της Λισαβόνας με σημαντική συμμετοχή στον τομέα της αλίας για την οικονομία της Γρυλανδίας και έχουμε τις επιπτώσεις για την κοινωνική ανάπτυξη και το περιβάλλον καθότι οι ακτικές ζώνες είναι ιδιαίτερως ευαίσθητες ε, για την κλωδία και την πανίδα τους. Οι αλληλευτικές δυνατότητες θα πρέπει επομένως να προσαρμοστούν προς τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο θα πρέπει να τηρεί ε, την διακήρυξη για την αστική αλληλεία ε, του Ιουλίου του 2015 που περιορίζει την αλία στον κεντρικό Αρκτικό ωκεανό για να διασφαλιστεί η διατήρηση του αρκτικού οικοστήματος. Το πρωτόκολλο που καλύπτει περίοδο 5 ετών προβλέπει χρηματική αντιπαροχή ύψους ε, άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το πρωτόκολλο πρέπει να ενισχύσει συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Ιλλανδίας για να προωθήσει την ανάπτυξη αηφόρου ελευτικής πολιτικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των ελευτικών πόρων στην ελευτική ζώνη της Ιλλανδίας. Πρόκειται για διάφορα είδη, όπως ο γάδος, το παλαϊκό κοκκινόψαρο, το πελαϊκό κοκκινόψαρο, υπόγλωσσα, γαρίδα ακτικής, καπελάνος και γραναδιέρος. Πρέπει να πριάγονται βιώσιμες ελευτικές πρακτικές για να διαφυλαχθεί η μακρόπνοη παραγωγικότητα της αλίας Κρυλανδίας και να στηριχθεί και η ελευτική πολιτική της χώρας αυτής. Το πλαίσιο αυτό η αδειοδότηση θα πρέπει να συνδεθεί στενότερα με το τοπικό εργατικό δυναμικό και τις τοπικές επιχειρήσεις το οποίο θα αυξήσει την αξία τη σχετική για την κοινωνική κοινωνία. Για την παροχή που συνδέεται με την ε, συμφωνία θα πρέπει να στηρίζει τη βιωσιμότητα του λευτικού του ομέα και να στηρίζει τη χώρα αναπτύσσοντα τι δυνατότητε τοπική απασχόληση ή στον τομέα τη αλληλεία. Και θεωρούμε ότι για αυτόν τον λόγο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου και ελπίζουμε να έχουμε και την στήριξη της ε, ε, Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος Τέλειου. Ευχαριστούμε και εμείς λέει η Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπέρ της τοποθέτησης του συναδέλφου για την αλληλευτική αυτή συμφωνία και θα έχει τη στήριξή μου για το νέο αυτό πρωτόκολλο που δείχνει τις στενές σχέσεις που έχουμε μεταξύ Αρακέσινου και Γρυλανδίας που όπως γνωρίζετε είναι ένα υπερατλαντικό υπερπόντιο μας το έδαφος όχι ευρωπαϊκό έδαφος θα μας επιτρέψει αυτή η συμφωνία να προαγάγουμε μια υπεύθυνη αλληλευτική πολιτική και βιώσιμη πολιτική αλληλεία για την Γλαδία και θα πρέπει να την επικυρώσουμε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ λέει πρόεδρο. Να πω απλώ ότι ο κύριος Φρανσούλη Κάζη έπρεπε να φύγει αλλά μου άφησε ένα σημείωμα που έλεγε ότι καθότι μπορούμε απλώς να συμφωνήσουμε ή να μην συμφωνήσουμε προτείνει να ακολουθήσει τον εισηγητή και να δώσει καταφατική απάντηση. Αυτά από την ομάδα των Σοσιαλιστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά την. Βεβαίω και έχετε δικαίωμα όπω και πριν, έτσι. Εννοείται αυτό πάντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλό απόγευμα. Πολύ σύντομα να πω απλώ ότι οι αρχέ τη νέα κοινή ελευθερικής πολιτική ε, αποτυπώνονται απολύτω καλά στο νέο πρωτόκολλο και αυτό ακόμα πιο συγκεκριμένα αποτυπώνεται στην συμφωνία με την Ιγλανδία για τις ε, ε, πλεονασματικές ε, αλλιευτικές δυνατότητες. Όλα αυτά είναι επικαιροποιημένα με τις τελευταίες επιστημονικές ενδείξεις και συμβουλές που έχουμε και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε αυτό για κάθε χρόνο διότι οι ποσοστώσεις που βλέπετε είναι ενδεικτικές και αιτήσιες. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας τις πιο πρόσφατες ενδείξει και στοιχεία. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι στο νέο αυτό πρωτόκολλο έχουμε αυξήσει κατά 10 με 15% την ούτως αποκαλούμενη τομεακή ενίσχυση που είναι αυτό το συστατικό της συμφωνίας που προσπαθεί να υποστηρίξει την τοπική αλληλεία του παρακτήου αυτού κράτους ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά μέγιστον τα 2,9 εκατομμύρια ενώ για την πρόσβαση πλέον με 13 περίπου εκατομμύρια και όλες οι ποσοστώσεις έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές σύμβουλες. Ευχαριστώ κατά τα άλλα τα μέλη της Επιτροπής για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την συνεργασία με τη Γενική Διευθυνσή σας, DG Mare. Έχετε τίποτε άλλο να πείτε, κάποια από εσάς. Τίποτε. Καλά. Προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών. Μια στιγμή να δω τη σημειώση μου. 27 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Εν προκειμένου μπορούμε μόνο να δεχθούμε ή να απορρίψουμε το πρωτόκολλο. Δεν μπορούμε δηλαδή να την τροποποιήσουμε. Ας το έχετε λοιπόν υπόψη και με τα λόγια αυτά σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Τελειώσαμε νωρί την συνεδριασία μα. Το επόμενο είναι question time, το υπαριθμό 10. Δεν έχουμε ερώτησεις, ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Έχω ωστόσο ένα μικρό αίτημα. Είδα στην ετήσια έκθεση του 2015 ε, αυτό το δημοσίευμα που ήρθε τα τέλη Νοεμβρίου είναι για την εξωτερική ε, πολιτική προς, προς, ε, προς τα έξω. Είναι ε, ε, ενδιαφέρον το κείμενο, έχει πολλούς πίνακες, είναι της έκθεση, έχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Απαντάει μέρη και σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοί μου προηγουμένως. Μου το έχετε ή τέλο πάντων το έχω εγώ, σε ασπρόμαυρο το αντίγραφο. Μήπως μπορείτε να το στείλετε εν χρωμό. Θα μας βοηθήσετε πολύ γιατί ορισμένοι από τους πίνακες είναι με χρώματα. Θα το διαβα... Ήμουν το διάβασα εγώ στο τρένο και τι μεγάλη χρησιμότητα έχει για μας. Το 11 είναι τα διάφορα, εάν κανείς έχει κάποιο διάφορο ε, να θέσει υπόψη μας. Στις 6.30 θα συναντηθούμε, υπενθυμίζω, με τους συναδέλφους μας της ε, βουλή των Κοινοτήτων. Θα μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσεις και αυτοί από μας. Και επανέρχεται λοιπόν στις 6.30 στην αίθουσα. Και μετά μπορούμε να ε, πιούμε και ένα ποτό μαζί τους. Στις 17 Φεβρουαρίου και στις 18, ολόκληρη 17 και το πρωί 18, θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Σας ξαναδώ στις 6.30.